So, Αγαπητοί συμμετέχοντες στη σημερινή μας συνάντηση, εργαστήριο, νομίζω ότι καλό μας έκανε αυτή η διακοπή για μεσημεριανό φαγητό. Είμαστε όμως, ελπίζω όλοι εδώ πάλι. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές και έχουμε και μια μικρή αλλαγή στο δεύτερο τμήμα. Ο μοναδικός άντρας που είχαμε εδώ δεν θα μπορέσει να έρθει. Θα το καταφέρουμε, καθώς και η κυρία Όμεν που θα αργήσει λίγο. Το θέμα αυτής της δεύτερης συζήτησης είναι οι συντάξεις, αλλά και η διαβίου κατάρτιση. Είναι ένα θέμα που σαφώς ε, μας αφορά όλους, αφορά άντρες και γυναίκες και Το θέμα είναι τι διαφορές υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των ανδρών και των γυναικών, αλλά και όταν φτάσουν στην ολοκλήρωσή της, στο τέλος, στην σύνταξη. Οι ομιλήτριες θα πάρουν το λόγο για πέντε λεπτά η καθεμία, για κάποια εισαγωγικά σχόλια. Εγώ στην πρώτη συζήτηση, κατά κάποιο τρόπο, έγινα αντιπαθής, γιατί είπα ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο ομιλίας. Το σκοπός μας είναι να γίνει πραγματικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων εδώ, γι' αυτό και σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτό το πεντάλεπτο. Α, ειδού και η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Καλώς ορίσατε. Η κυρία ο Μεν Ρόιτεν είναι Ολλανδέζα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αρμόδια για θέματα απασχόλησης. Έχει υποβάλει νομοθετικά κείμενα, ψηφίσματα και όπως ε, όλοι παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν κοινωνικά θέματα που εμπλέκονται και ε, σε πολλά άλλα βεβαίως ε, θέματα εμπλέκονται τα κοινωνικά θέματα. Αριστερά μου βρίσκεται η κυρία Ματέρα από την Ιταλία, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και αρμόδια για τη γνωμοδότηση της ε, αρμόδιας αυτής της Επιτροπής για την έκθεση της κυρίας Όμεν Ρόιτεν. Η κυρία Έμτζεν. Μου είχε δώσει ένα κείμενο το οποίο το έχασα, ένα κείμενο που έπρεπε να το διαβάσω εκπροσωπεί τους ε, εργαζόμενους, τους ε, εργοδότες. Θα ακούσουμε διαφορετικές ε, απόψεις και εκτιμήσεις και βεβαίως είναι εδώ και επικεφαλής της ε, αρμόδιας ομάδας που ασχολείται με θέματα απασχολησιμότητας γυναικών συντάξεων. Επίσης, ε, Business Europe, Business Europe είναι μια ομάδα εργασίας ε, για την κοινωνική προστασία και εκπροσωπείται από την πρόεδρο Λος Βαν Έντεν. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν θα ξεκινήσει με την παρουσίασή της για πέντε λεπτά. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, γιατί αν ο καθένας από μας σαν Ευρωβουλευτής δεν μιλήσει τη γλώσσα του, τότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν πρόκειται να το κάνει για μας. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί μπορεί να αναφέρω και κάποια πράγματα στα αγγλικά. Θα μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κάθε φορά που έχουμε επισκέπτες εδώ, λέω ότι αν η Ευρώπη δεν είχε κάνει τίποτα, σήμερα θα υποφέραμε από το Ολλανδικό σύστημα. Η Λούς με γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια από τότε που ήμουν μέλος του Ολλανδικού Κοινοβουλίου τότε που οι γυναίκες ε, πολέμησαν για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες. Πολλές ε, δράσεις ξεκίνησαν και μας οδήγησαν σήμερα σε αυτή την ίση μεταχείριση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορές στις αποδοχές. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε γρήγορα το πρόβλημα αυτό σήμερα. Μία γυναίκα στις 5 μπορεί να πέσει στην χαμηλότερη μισθολογική κατηγορία είτε να πληγεί από την φτώχεια. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς επειδή κάνουμε παιδιά, διακόπτεται η επαγγελματική μας στρατιοδρομία, είναι όλο και πιο δύσκολο να συγκεράσει κανείς ε, την επαγγελματική του και την οικογενειακή του ζωή. Πολλοί προσπαθούν να εργαστούν από το σπίτι με αποτέλεσμα οι γυναίκες να έχουν λιγότερες δυνατότητες ε, να κερδίσουν αξιοπρεπείς μισθούς. Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Και αυτό που προσπαθώ να καταλάβω τώρα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Ήμουν εισηγήτρια για την πράσινη βίβλο Και βεβαίως ε, τώρα διαπιστώνουμε ότι η νομοθεσία μεν υπάρχει, αλλά δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα έτσι να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εγώ μιλούσα με τους συνεργάτες μου πριν από λίγο και διαπίστωσα ότι το θέμα της ισότητας των αμοιβών των μισθών είναι ένα κεντρικό θέμα. Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει μία σειρά προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μου πείτε ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άντρες, η απάντηση είναι πολλές φορές ότι θα πρέπει να αναλάβουν το θέμα αυτό οι εργοδότες. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης θα ήταν μια λύση. Οι γυναίκες που εργάζονται σε χαμηλότερες ε, μισθολογικές ε, κατηγορίες θα πρέπει επίσης να δουν μια αναβάθμιση των ε, μισθών τους. Στην Ευρώπη μπορούμε βεβαίως να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να καθορίσουμε το γενικό πλαίσιο, της κατευθυντήριας γραμμές, τα κράτη-μέλη όμως καλούνται εδώ να δραστηριοποιηθούν. Η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, επαναλαμβάνω, αλλά και μέτρα συνοδευτικά έτσι ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να συνδυάσουν την οικογενειακή και προσωπική του ζωή με το επαγγελματικό τους ε, ε, σχέδιο, με το επάγγελμά τους. Το θέμα των συντάξεων. Σε 10 χρόνια δύο εργαζόμενοι θα στηρίζουν και θα τροφοδοτούν την σύνταξη ενός συνταξιούχου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εργαζομένους, άρα περισσότερες γυναίκες. Υπάρχουν κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση των ε, γυναικών και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει σαφώς να κάνουμε κάτι έτσι ώστε οι γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας και να παραμείνουν και έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν με ικανοποιητικό τρόπο οι συντάξεις. Ελπίζω ότι οι νέοι δεν θα συνεχίσουν να εθελοτυφλούν. Θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταφραστούν σε λόγια αυτές ε, οι, ε, σε πράξεις αυτές οι ωραίες προτάσεις. Σας ακούω να είστε πολύ θετικοί και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι και θετικοί. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ε, Κυρία Ματέρα, Μπάρβαρα Ματέρα. Sì, buongiorno a Θα ήθελα όλους τους συναδέλφους να τους ε, ευχαριστήσω. Λυπάμαι που δεν ήρθε εδώ ο συνάδελφος Νταρντέν, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψη ενός ε, συναδέλφου ανδρός και τέλο πάντων θα πρέπει να τηρήσω το χρονικό όριο το οποίο είπε η κυρία Κοχμέρη. Και στην Ιταλία δεν τα πάμε τόσο καλά όσον αφορά τέτοιου είδου ε, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία Τέλο πάντων θα προσπαθήσω να κινηθώ σε αυτά τα πλαίσια και ευχαριστώ πρώτα από τη Γενική Διεύθυνση τη Επικοινωνία του Κοινοβουλίου που οργάνωσε αυτή την ημερίδα που ε, ε, αφορά ακριβώ την γεφύρωση του μισθολογικού χάσματο. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το ότι όλα αυτά γίνονται και έχουμε την ευκαιρία της 8ης ε, Μαρτίου. Α, τα, τα λέω πάρα πολύ, δεν προσθέτω να μεταφράσετε. Καλά, καλά. Λοιπόν, μιλούσαμε για το μυστορικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο αφορά μια δυσμενή διάκριση πάρα πολύ σημαντική και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, πλήστε γυναίκε παντού. 17,7% είναι ο μέσο όρο ε, αυτού του χάσματο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, 5% σε κάποιε χώρε όπω η Ιταλία και όμω το μάξιμο είναι 30% σε κάποιε χώρε όπω η Εστονία. Πρόκειται για αυτό το χάσμα λοιπόν το οποίο ε, επιφέρει πάρα πολύ σημαντικέ συνέπειε όσον αφορά ε, τον υπολογισμό τη σύνταξη όταν έρθει η ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι οι γυναίκε έχουν προσδόκιμο ζωή μεγαλύτερο, καλύτερο τέλο πάντων από του άντρε. Οπότε εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει εδώ ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν σε κατάσταση φτώχεια οι, οι, οι γυναίκε, 20% των γυναικών ε, πάνω από τα 65 χρόνια ε, είναι ευάλωτες σε αυτό το φαινόμενο δηλαδή του να πέσουν σε, σε, κατάσταση παινίας φτώχειας. Το Δεκέμβριο του 2010 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτού του είδους τα προβλήματα στην πράσινη βίβλο που αφορά την, την, την ισότητα των φύλων. Να προσέξουμε επομένω ε, το θέμα των συντάξεων. Κυρία Όμιν Ράιτον ασχολήθηκε και εκείνη. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάσει τι σχετικέ βασικέ γραμμέ, των προσανατολισμού. Και είχα την ε, τιμή και εγώ να ε, αναλάβω μια σχετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων Γυναικών και της Ισότητας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο στόχο μα, στα πλαίσια αυτή τη εκθέση ήταν να τονίσουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η ανισότητα και από πλευρά συντάξεων. Στα πλαίσια λοιπόν τη ε, ενασχόλησή μου με αυτή την ε, έκθεση είπαμε ότι είναι πάρα πολλέ αυτέ οι γυναίκε, οι οποίε αδικούνται και όσον αφορά το συνταξιδοτικό. Ε, πολλές φορές οι γυναίκες ε, διακόπτουν την ε, επαγγελματική του αδειοδρομία για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Μιλούμε για τις υποχρεώσεις. Αυτό είναι μια δυσμενής διάκριση. Και καταλήγουν επομένως να έχουν σύνταξη μικρότερη από τους άνδρες. Αυτό, επομένως, τις κάνει ακόμη πιο ευάλωτες στον κίνδυνο του να πέσουν σε κατάσταση παινίας. κυρία Μπάουερ ήρθε και εκείνη ασχολήθηκε με το πρόβλημα και προωθήσαμε μια σειρά πρωτοβουλειών. Το Κοινοβούλιο βεβαίως και πρέπει να αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Πάρα πολύ είναι ο χρόνος που αφαιρούν οι γυναίκες στις οικογένειε στα παιδιά που έχουν και επομένως αυτό έχει τις επιπτώσεις που προαναφέραμε στον υπολογισμό της σύνταξης. Είμαι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι πάρα πολύ σωστά η Επιτροπή ξεκίνησε αυτή την ευρεία δημόσια διαβούλευση. Ούτω ώστε να δούμε ποια θα είναι τα στοιχεία που πρέπει να καλύψει η λευκή βίβλος που θα αφορά το συνταξιοδοτικό. από τις πρώτες μέρες της ε, διαβούλευσης πήραμε χιλιάδες απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια. Ένα σωρό απόψεις που θα τις καλύψουμε στην ε, Λευκή Βίβλο. Αυτή η Λευκή Βίβλος δημοσιεύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του εναστότος έτους και επίσης προτείνονται εκεί μέτρα για τον αρμονικό συνδυασμό του οικογενειακού με τον επαγγελματικό βίο. Επίσης είπαμε ότι έτσι θα προχωρήσουμε προς την γεφύρωση του χάσματος. Τα ηλικιακά όρια, όλα αυτά πρέπει να αφιγραμμιστούν, να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Το 2020 Να σταματώ, σταματώ κάθε τόσο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να κάνω αυτές τις μικρές πάυσεις, τόσο ώστε να μπορούν οι διερμηνείς να προλάβουν να μεταφράσουν αυτό το οποίο λέω. non ho sforato. Sto per concludere. Πάρτε, πάρτε μια ανάσα και συνεχίζουμε. A little bit? Oh, you need more time? No, no, no, no, no. Okay. Only one minute. Nell'Unione Europea... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγα. Να, να, να. Πήραν μία, δύο ανάσες και παραπάνω. Λοιπόν, Έχουμε, θα, θα είμαστε λοιπόν 28, 28 μέλη το 2020 και θα πρέπει τότε να φεγανιστούν τα στεξιωτικά όρια. Θα πρέπει να πάρουμε κάποια αποτελεσματικά μέτρα, ούτω ώστε να μπορούν οι γυναίκε να εργάζονται όσο μπορούν καλύτερα την ώρα που θα πάρουν τη σύνταξη, να έχουν κάποια οικονομική σύνταξη όπω οι άντρε. Τώρα, ε, εν είδη συμπερασμάτων λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι θέλουμε να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να είναι βιώσιμα, θα πρέπει κάποια κριτήρια τα οποία να εξασφαλίζουν την ισότητα της μεταχείρισης και έτσι να αποφύγουμε το να, να, πρέπει να βρίσκονται προ κάποιες δύσκολες επιλογές οι γυναίκες μεταξύ δηλαδή οικογένειας ή, ή σταδιοδρομίας. Ε, θεωρώ επομένω ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν ε, προοδευτικά να προσαρμόσουν τη μία δραστηριότητα με την άλλη. Πρόκειται επομένω, για, για αγώνες που πρέπει να δοθούν, δίνονται καθημερινά εδώ στο Κοινοβούλιο και επομένως ε, όλοι όσοι ε, θέλουν θα, θα, πρέπει να βοηθήσουν και σε επίπεδο κρατών μελών τόσο ώστε να προωθηθεί η υπόθεση των δικαιωμάτων τη γυναίκα. Γιατί, α πούμε, πολλέ φορέ τίθεται το ερώτημα γιατί ένα άνδρα να είναι μέλο τη Επιτροπή των Γυναικών, διότι εδώ αυτό είναι θέμα δικαιωμάτων, θέμα ισότητα. Επίσης, αυτά που σας είπα στην αρχή της ε, εισήγησής μου, δυστυχώς, ισχύουν. Οι γυναίκες είμαστε δυστυχώς ακόμα θύματα δυσμενών διακρίσεων και στον χώρο της δουλειάς. Επομένω θα πρέπει και αυτό το πρόβλημα να ακολουθήσει την υπόλοιπη πρόοδο που έχει σημειώσει η κοινωνία μας. Αυτά. Από ό,τι βλέπω τελείωσε ο χρόνο μου και σα ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ παθιασμένη σας παρουσίαση, τη δέσμευσή σας. Ε, ζητήσατε ένα λεπτό, ένα λεπτό όμως πολιτικό λεπτό, έτσι. Δεν σπάω, αστείευομαι. Πρόκειται λοιπόν για θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους, που μας αφορούν όλους. Τώρα θα περάσουμε από την πολιτική στην οικονομία. Κυρία Άντερς, Business Europe. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ την οργάνωση Business Europe αλλά μιλώ με την ιδιότητα της Ολλανδής εκπροσώπου του Συλλόγου Εργοδοτών Θα μιλήσω Ολλανδικά για να δείξω εμφανώ αλληλέγγυα προς την κυρία Όμεν Ρόιτεν. Μπορείτε να φανταστείτε σίγουρα ότι η Business Europe προάγει ε, τα ζητήματα ισότητας ε, των δύο φύλων. Ε, δεν συμφωνούμε απλώς με την αρχή, την έννοια δηλαδή της ισότητας, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η αρχή στην πράξη και τα μέλη του Business Europe καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της ισότητας. Όταν συζητούμε για τα, τις ε, διαφορές στη μεταχείριση ανδρών και γυναικών ε, και το μισθολογικό χάσμα που χωρίζει τα δύο φύλλα, έχουμε ε, μία μάλλον συλλογική εικόνα της κατάστασης, δηλαδή εξετάζουμε ποιος είναι ο μέσος μισθός ενός άντρα σε μία χώρα ε, ή ποιες είναι οι μέσες αποδοχές της γυναίκας στη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, ε, ανάγεται σε συλλογικό θέμα αν θέλετε και δεν εξετάζεται η ίδια η διακριτική μεταχείριση. Ε, το μισθολογικό χάσμα είναι φυσικά ε, κάτι που πρέπει να καταπολεμήσουμε, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα ε, υπό μια διαφορετική οπτική γωνία και όχι αυτή της διακριτικής μεταχείρισης, κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να σχολιάσω εντάχει Ε, τις αιτίες αυτής της ε, συλλογικής, ε, μαζικής μάλλον, μισθολογικής διαφοράς. σωστά ε, αναφερθήκαμε στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, ε, αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος ε, παράγοντας, ο μόνος καταλητικός παράγοντας. Εξαρτάται από το αν θέλει κάποιος να απασχοληθεί πλήρως ή μερικώς, πόση ευελιξία θέλει σε σχέση με την αιτήσια άδεια και ούτω καθεξής. Όταν εξετάζουμε ε, την σχέση τώρα ανάμεσα στην, ε, στο μυθολογικό αυτό χάσμα και την ε, διαφορά ως προς τις συντάξεις. Συνειδητοποιούμε ότι ε, δεν θα μπορούσαν ε, πάντοτε να αποδοθούν σε ε, λόγους διακριτικής μεταχείρισης. Θα μπορούσαμε όμως φορές να αποδώσουμε αυτές τις διαφορές στην αγορά εργασίες στη μορφή που έχει σε κάθε χώρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπομισθούν τις δικές τους ευθύνες και εξάλλου θα είναι υποφελές όχι μόνο για τις ε, άμεσα ενδιαφερόμενες, αλλά και για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα ε, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα των ε, κρατών μέλων. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω την προσοχή μου σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την συνταξιοδότηση. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης ε, ε, διαφέρει για τα δύο φύλλα. Αυτό νομίζω εδώ θα πρέπει να ρυθμιστεί. Εάν θέλετε όλα τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα όλα τα ταξιδιωτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, ευθυγραμμιστούν, ε, τελικά νομίζω ότι θα αυξηθεί το ηλικιακό όριο ταξιοδότηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί μια λύση από όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, εάν ασχοληθούμε ε, με τα ωφέλη που αποκομίζει κανείς από τα επικουρικά συνταξιοδοτικά συστήματα, συνειδητοποιούμε ότι ε, υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες ε, έχουν χαμηλότερες αποδοχές ούτως ή άλλως από τους άντρες διότι επιλέγουν διαφορετικού είδους σταδιοδρομίες, απασχολούνται μερικώς ή ζητούν παρατεταμένες άδειες άνευ αποδοχών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Οι ασφαλιστικές εισφορές και η κατοχήρωση των συντάξιμων ε, χρόνων και των ε, συντάξιμων δικαιωμάτων, κυρίως για τις επικουρικές συντάξεις, ε, συνδέονται με το εισόδημά σας, με το μισθό σας. Εάν δεν έχετε αποδοχές, δεν μπορείτε να συνεισφέρεται παρκώς στα ασφαλιστικά συστήματα και άρα ε, θα έχετε μειωμένη σύνταξη. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας κανόνας που ισχύει γενικά και πρέπει όλοι να τον αποδεχτούν. Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί επίσης ε, για ποιο λόγο οι άνθρωποι ε, τίνουν να ζητούν παρατεταμένες ε, γονικές άδειες, ε, ορισμένες φορές ε, άνευ αποδοχών, άλλες φορές παίρνουν τη μορφή επιδομάτων πρόνοιας, άλλες περίοδοι δεν είναι μεν ένα άνευ αποδοχών, αλλά μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από πλευράς του ερωδότη. Ε, υπάρχουν ε, κοινωνικοί εταίροι σε κάποια κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, στις συζητήσεις σχετικά με την αναμόρφωση των συνδεξιδοτικών συστημάτων. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο να βρούμε ε, τις πιο πρόσφορες για κάθε χώρα λύση. Θα τελειώσω με ένα παράδειγμα από την Ολλανδία, ε, όπου ισχύει μία συλλογική συμφωνία, δηλαδή δημιουργήθηκε η δυνατότητα για μία αυστηρός προσδιορισμένη χρονική περίοδο να ε, παίρνει κάποιος άδεια άνευ αποδοχών, αλλά συνεχίζει, να συνεχίζει συγγνώμη, να καταβάλει ε, τις ασφαλιστικές του εισφορές. Αλλά αυτό φυσικά λειτουργεί σε θελοντική βάση. Έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, ε, θα ακούσω καλύτερα τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Και Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα μπορέσουμε βεβαίως να εμβαθύνουμε κάποια σημεία που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. Ωραία. Λοιπόν, εξ ονόματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα δώσουμε το λόγο σε κάποιον που ήταν ε, εργαζόμενοι στην Όπελ, στο Βερολίνο, Θα μιλήσω γερμανικά. Πριν μιλήσω για τις επιχειρήσεις και για τα θέματα που αφορούν άμεσα το θέμα που μας αφορά, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις συντάξεις και όσον αφορά τα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα, βλέπουμε πάρα πολλά θετικά σημεία και προτάσεις στην ε, Λευκή Βίβλο. Οι διαφορές ε, που φαίνεται να συνεχίσουν να υπάρχουν μεταξύ των συντάξεων και των ε, διαφόρων προϋποθέσεων για να φτάσει κανείς στη σύνταξη μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που έχει φυσικά τραβήξει την προσοχή ε, πολλών κρατών μελών, αλλά και πλέον συζητείται ευρέως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση σε αυτή τη λευκή βίβλο αναφέρεται στις δυνατότητες να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση των συντάξεων, λέγοντας βεβαίως ότι αυτό δεν είναι η μόνη λύση υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες, κάποια άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να υπάρξει πιο ίση μεταχείριση μεταξύ των ανδρών και των γυναικών που φτάνουν στο όριο ε, συνταξιοδότηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να δούμε το μέσο όρο και αυτό που γενικώ ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικές γραμμές οι αριθμοί που βλέπουμε είναι ένα 50% χαμηλότερες συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο Λουξεμβούργο παραδείγματος χάρη. Αλλά και σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφορετική οικογενειακή πολιτική και τα διαφορετικά συνοδευτικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί στις χώρες μέλη και που οδηγούν σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές και ανισότητες. Υπάρχουν λοιπόν χώρες όπου οι διαφορές αυτές είναι εξαιρετικά εντυπωσιακέ. Είναι θέμα βεβαίως, όπως σας είπα, και γενικότερης πολιτικής. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τη γενικότερη πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της οικογενειακής ε, ε, πολιτικής. Σίγουρα ε, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα τα οποία αν θέλετε μπορώ να σας τα παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιο δίκαιη κατάσταση. Η πρώτη όμως κατεύθυνση θα πρέπει να είναι βεβαίως το ίδιο, ε, ίδια ηλικία συνταξιοδότησης για άντρες και γυναίκες, κάτι που βεβαίως θα οδηγήσει ε, στην ε, επιμήκυνση της ε, επαγγελματικής ζωής. Υπάρχουν κλάδοι που βεβαίως ο αριθμός των ανδρών είναι πολύ μεγαλύτερος και εκεί βλέπουμε οι διαφορές να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακές. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση για τις γυναίκες σε αυτούς τους κλάδους, σε αυτούς τους τομείς, όπως τη βιομηχανία, στους ε, κλάδους αυτούς βεβαίως υπάρχουν πολλές φορές ε, και κάποια ειδικά καθεστώτα που διέπουν ε, τις συντάξεις, όπως παραδείγματος χάρη συγκεκριμένες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Ε, επίσης, σε εθνικό επίπεδο διαπιστώνουμε ότι πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Όσον τον τρίτο πυλώνα που είναι η ιδιωτική ασφάλιση, είτε πρόκειται για ασφάλεια ζωή, είτε για άλλου είδους ε, επικουρικές συμβάσεις ή άλλου είδους επιδόματα. Ε, από ό,τι φαίνεται από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη επεξεργασία και εδώ οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερες αποδοχές και βλέπουμε ότι σε κάποιες ειδικέ μισθολογικές κατηγορίες οι συντάξεις αυτές είναι πραγματικά ελάχιστες για τις γυναίκες. Σήμερα το οικογενειακό μοντέλο είναι πολύ πιο ευρύ και πολύμορφο θα έλεγα σε σχέση με το πώς ήταν η οικογένεια πριν από 30 χρόνια. Αυτό και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε διάφορες προσαρμογές. Σήμερα βλέπουμε ότι πολλές ε, πολιτικές οδηγούν σε αυτές τις διαφορές μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο φυσικά θα πρέπει να το εξισορροπήσουμε, να γεφυρώσουμε το χάσμα. Αλλά βεβαίως αν θέλετε μου να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες ε, σε συγκεκριμένα θέματα που σας αφορούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε ακριβώς πέντε λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες προοπτικές για ένα πρόβλημα το οποίο όλοι έχουμε εντοπίσει σαν πρόβλημα παρόν σε όλες τις χώρες μέλη. Ακούσαμε τις απόψεις των μεν και των δε την άποψη, αν θέλετε, των ε, νομοθετικών ε, αρχών, των ε, κοινωνικών εταίρων, αλλά και των συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων. Υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν παρατηρήσεις που θα θέλετε να κάνετε σε αυτό το σημείο. Είναι ένα θέμα που ίσως ε, μπορεί να σας φανεί τεχνικό. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι είναι κάτι που θα απασχολήσει τον καθένα από μας. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν παρουσίασε πολύ σωστά αυτήν την, ε, αν θέλετε, κατάσταση που όλοι θα αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας και το γιατί τα αποτελέσματα φαίνονται τόσο διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη. Γιατί η αγορά εργασίας είναι διαφορετική. Η παρουσία και η πρόσβαση των γυναικών είναι διαφορετική. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα δυνατότητας χρηματοδότησης. Εδώ είναι θέμα σύγκρουσης γενεών. Οπότε και τα συνδικάτα θα πρέπει πάρα πολύ προσθετικά να το σκεφτούν. Οι εργαζόμενοι να κάτσουν για να σκεφτούν τι θέλουν για τα παιδιά τους. Θέλουν να μην μπορούν πια τα παιδιά τους να κάνουν οικογένεια μια που το κόστος θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και πάλι το θέμα του ορίου συνταξιοδότησης και να δούμε πώς μπορεί αυτό να συγκεραστεί καλύτερα. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ευτυχώς πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι ακόμα έχουν το δυναμισμό των νιάτων αλλά θα πρέπει όλο ένα και περισσότερους να καλύψουμε όλο ένα και περισσότερους δηλαδή μπαίνουν σε και μένουν δηλαδή δουλεύουν περισσότερα χρόνια ένα αυτό το άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να μάθουμε ότι κανείς θα πρέπει να αποταμιεύει για την σύνταξή του. Να βάζει δηλαδή χρήματα στην πάντα. Αυτά οι διάφορες μορφές συντάξεων να καλυφθούν. δω να κάποιο ούτε να θέλει να ανέβει το στεξιωτικό όριο, ούτε να δουλεύει περισσότερο. Ε, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει μας οι κοινωνικοί εταίροι να κάτσουν, να σκεφτούν και να αποφασίζουν. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ λογικό κάποιο στην ηλικία των 68 ξαφνικά να λέει ότι να πάμε στα 65 το όριο, ενώ το, το προσδόκιμα ζωή μπορεί να έχει φτάσει ας πούμε, στη δική μου χώρα, στις κάτω χώρες, δηλαδή στα 80. Άρα δεν θέλουμε ούτε να έχουμε καμία κλιμάκωση αυτού του χάσματος και σύγκρουση γενναιών. Η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση. Έχετε το λόγο. Το ερώτημά μου είναι αν ε, το θέμα του ορίου συνταξιοδότησης της ηλικίας τι ακριβώς είναι η πρότασή σας γιατί σε εμά στην Αυστρία είναι 60 για τι και 65 για του άντρε. Ζητάτε ίσιο ίδιο όριο ηλικίας. Κοιτάξτε, ναι, αλλά αυτό δεν το προτείνω για να επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που δεν είναι λόγο δεν έχω καμία πρόθεση να σας επιβάλλω ή να σας πω αυτό πρέπει να επιβληθεί ή το άλλο. Είναι δικό σας θέμα, δική σας επιλογή. Αλλά σίγουρα θα οδηγηθούμε σε περισσότερη εργασία, περισσότερα χρόνια και επιμήκυνση του επαγγελματικού βίου. Το ερώτημα είναι αν όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που ισχύει σήμερα. Όσον αφορά την πράσινη βίβλο, είδατε ποιες είναι οι προτάσεις. Κυρία Μπάουερ. Μπάουερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως θα ενδιαφέρον σήμερα η Eurostat σήμερα να κοινοποιήσει αυτό το οποίο θέλει να δημοσιεύσει την 8η Μαρτίου. Γιατί τα στοιχεία εκείνα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ο τίτλος είναι 40% περισσότερες γυναίκες παρά άντρες είναι πάνω από 65 ε, στην, στην, στην Ευρωπαϊκή Δηλαδή, ε, διαφορά 40%. Τι πάει να πει αυτό, ότι έχουμε πολύ περισσότερες γυναίκες έχουμε ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και 40% είναι εντυπωσιακό, είναι τρομερό κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό έχουμε 62 εκατομμύρια γυναίκες που κινδυνεύουν να πέσουν σε κατάσταση φτώχειας. Και 50 εκατομμύρια άντρες, δηλαδή 8 εκατομμύρια διαφορά δεν είναι και λίγο. Σας ευχαριστώ. Αυτά απλώ ήθελα να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Αυτό αναδεικνύει κάποια θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα στατιστικά στοιχεία και συγκρίσιμα στοιχεία και τις πληροφορίες έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και έτσι ώστε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την ισότητα των φύλων, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες να μπορέσει να φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιόπιστα. Τώρα, όσον αφορά το όριο συνταξιοδότησης, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. 30-35 χρόνια είναι ο μέσος όρος μιας επαγγελματικής ζωής, αλλά το 46% των εργαζόμενων δεν φτάνουν καν στο παρόν υπάρχουν και ισχύον όριο συνταξιοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, να φτάνουν μέχρι αυτό το όριο συνταξιοδότησης, την ηλικία συνταξιοδότησης και να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες θα επιτρέψουν σε όλους όσους έχουν φτάσει σε αυτό το όριο κατόπιν βεβαίως να έχουν μια ε, ίση σύνταξη. Το θέμα είναι ότι το αν θα επιμηκυνθεί ή όχι η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής εξαρτάται από πολλά άλλα θέματα. Είδαμε παραδείγματο χάρη ότι η διαρκεια της επαγγελματικης ζωης εξαρταται απο πολλα αλλα θεματα ειδαμε παραδειγματος χαρη οτι η νέοι ξεκινάνε όλο και πιο αργά την εργασία τους. Μπαίνουν στην επαγγελματική ζωή στα 25, στα 30. Καταλαβαίνετε, στην Ισπανία ας πούμε έχουμε το μέσο όρο 25. Καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει κανείς στα 30-35 ε, χρόνια επαγγελματικής ε, σταδιαδρομίας σίγουρα θα πρέπει να ξεπεραστεί πολλές φορές το όριο συνταξιοδότηση και το θέμα της ανεργίας. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό επιβραδύνει την ολοκλήρωση της επαγγελματικής ζωής. Εμάς όμως, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι συνθήκες εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική μελέτη, την οποία έχουν συνεισφέρει Βεβαίως και οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Η κατάσταση δείχνει ότι βάσει αυτής της μελέτης 25 με 30% των εργοδοτών επιθυμούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση των συνθήκων εργασίας με πολύ συγκεκριμένες μέτρες. Ιδιαίτερα με την απασχόληση και μεγαλύτερων εργαζομένων, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων. Δίνοντας ε, δηλαδή τη δυνατότητα σε έμπειρους, ε, πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να παραμείνουν στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται σαν τάση οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν και θα πρέπει να αποκτήσουν και περισσότερες ε, ευκαιρίες και δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, μπορείτε να το δείτε. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Τρεις ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις θα κάνω μόνο. Μπάρμπαρα, ένα λεπτάκι. Ε, μας λένε ότι θα πρέπει να συνταξιοδοτούνται στην ίδια ηλικία οι άντρες με τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν ε, συμφωνώ εγώ με αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παραμένουν για ε, μακρύτερο χρόνο στην αγορά εργασία. Ε, οι γυναίκες, αλλά ξέρετε δεν είναι εξίσου σοβαρά τα προβλήματα σε όλε τι χώρε. Αν, ε, κοιτάξτε. Ωραία. Κάνατε και τις σα παρατήρηση. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα που ακούσαμε προηγουμένως, δηλαδή αν είμαστε υπέρ ή κατά τη ευθυγράμμιση της ε, ταξιοδότηση ε, των ανδρών και των γυναικών. Αν αυτό θα επιτρέψει να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρόνο ε, στην αγορά εργασίας οι γυναίκες. Εξαρτάται από τη χώρα θα σας απαντήσω. Ε, αυτό σημαίνει βεβαίω ότι οι άντρε θα πρέπει να επομεστούν τις ευθύνες του σε άλλους τομεί. Ε, ε, η εκπρόσωπος του Business Europe αναφέρθηκε στο θέμα της άδειας της γονικής άδειας, της άδειας μητρότητας. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη της άδειας πατρότητας. Δηλαδή αναφέρεται π.χ. στην Ιταλία η άδεια πατρότητας, αλλά ε, δεν λειτουργεί το σύστημα. Πάντως είναι θέμα ανάληψη ε, ευθυνών από πλευρά ε, των ανδρών στις λεγόμενες βόρειε χώρες. Είναι πρωτοπόροι οι άντρε κατά τη διαστολή με τους ουραγούς όπως είναι οι Ιταλοί άντρες παραδείγματος χάρη σε θέματα διασπατρότητας ε, θα πρέπει να σεβόμαστε τις οικογενειακές ευθύνε των γυναικών. Μιλήσαμε για στα σταδιοδρομίες ε, των γυναικών, διότι πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους. Ε, νομίζω ότι αυτή η περίοδος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μία περίοδο ασφαλιστικών εισφορών, τόσο ώστε να κατοχυρώνεται η σύνταξη. Ναι, λοιπόν, απαντώ υπό κάποιους όρου. Ευχαριστώ. Κάποιοι άντρε εδώ. θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που ακούσαμε. Ε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, ως προς την ε, ίση μεταχείριση υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές και για τις βασικές και για τις επικουρικές συντάξεις. Είπατε κι εσείς ότι το 90 ε, εξέδωσε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο που προβλεπόταν ότι είναι παράνομη οποιαδήποτε μισθολογική διαφορά ανάμεσα ε, στις γυναίκες και τους άντρες. Νομίζω είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε. Τώρα, ως προς ε, τα συνδικάτα εργαζομένων θα μπορούσα να σας πω ότι ένα το επιχείρημα ότι κάποιοι δεν φτάνουν μέχρι το όριο συνταξιοδότησης και χρησιμοποιούν κάποιοι αυτό το επιχείρημα για να αυξήσουν το όριο συνταξιοδότησης ε, δεν ευσταθεί, γιατί όντως κάποιοι δεν φτάνουν ποτέ σε αυτήν την ηλικία. Αλλά εάν αυξηθεί μέσω νόμου ε, το όριο συνταξιοδότησης, θα επηρεαστεί η πραγματική επαγγελματική ζωή των ασφαλισμένων. Μας μιλήσατε επίσης για τους ε, ηλικιωμένους, την απασχόληση των πιο ηλικιωμένων. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ε, το τωρινό σύστημα δεν λειτουργεί εύρυθμα και έχουν ήδη γίνει προσπάθειες ε, για να αλλάξει η νοοτροπία των εργοδοτών ούτω ώστε σε μια προχωρημένη, πιο προχωρημένη ηλικία να μπορούν ε, οι άνθρωποι να βρουν μια θέση εργασίας. Κάναμε μια μελέτη για αυτό το θέμα και έχουμε μοιράσει τα αποτελέσματα στα μέλη του Business Europe. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω από την Ισπανία είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι, για την κυρία Ματέρα, μια ερώτηση μας ε, ανέφερε για το κατά πόσον ε, θεωρείται ή μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ε, η αποδοσίωση στα παιδιά ή η ενασχόληση τα παιδιά σαν κομμάτι της σύνταξης. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, αυτό μου φαίνεται λίγο ουτοπικό. Τέλος πάντων, εσείς τι λέτε, τι, τι, πιθανότητες υπάρχουν αυτό, το, αυτή η ιδέα να προωθηθεί, ματέρα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, ίσως τώρα ακούγεται αυτό λίγο ουτοπικό αυτή η πρότασή μας, αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως και είπαμε ότι συζητήθηκε στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών πριν από λίγους μήνες και το ξέρουν αυτοί οι συνάδελφοι. Είχαμε εκπροσώπους από διάφορα κράτη-μέλη. Ναι. Ίσως αν ξεκινήσει αυτή η από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως θα μπορεί, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με αυτό, να δούμε δηλαδή πώς αυξάνεται η εξάρτησή μα από τα συντηρητικά συστήματα. Πάντω, εν πάση πρόκειται για μια πρωτοβουλία πάρα πολύ θαραλέα. Είναι ένα όνειρο, ένα όραμα. Εμείς, ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων, ίσως μια μέρα δούμε αυτό το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Πολύ σωστά τα είπατε. Η σημερινή συγκυρία, κάτι κράτη-μέλη, δεν επιτρέπει σήμερα μια τέτοια πρωτοβουλία να πιάσει τόπο. Όμως εδώ στο Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη. Πρόεδρος. Ναι. Μπορώ να στηρίξω αυτή την πρόταση, σαφώς, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε αυτά τα συστήματα. Είναι βεβαίως πολύ πιο εύκολο να βρει κάποιος τέτοιες δυνατότητες από τα δημόσια συστήματα συνταξιοδότηση τον ιδιωτικό τομέα και οι επιχειρησιακές ε, συντάξεις δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες. μερινά από λίγα χρόνια είχαμε δει ότι υπήρχαν δυνατότητες για μια γυναίκα να υπολογίσει το ποσό της σύνταξής της βασιζόμενη στο μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών τριών, ε, ή των τριών ετών ε, με την υψηλότερη μισθοδοσία. Ο υπολογισμός ε, αυτός γινόταν επίσης και για το εφάπαξ που έπαιρναν οι γυναίκες. Και εκεί βεβαίως ε, όταν και ο αριθμός των παιδιών που είχαν οι γυναίκες, το κατά πόσο είχαν πάρει η μητρική άδεια ή όχι, τη διάρκεια. Υπάρχουν γυναίκες που αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι 10-15 χρόνια ε, για οικογενειακούς λόγους. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Σαφώς και υπάρχουν περίπλοκες τεχνικές λεπτομέρειες. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι συγκρίσιμες οι καταστάσεις από τη μια χώρα στην άλλη. Έχετε το λόγο, απλώς πείτε πολύ σύντομα ποιος είστε. Κάθριν Χάκετ από το κέντρο ε, ερευνών στο Λονδίνο. Θα ήθελα να ρωτήσω Σε σχέση με αυτήν την πολύ προχωρημένη και προοδευτική και τολμηρή πρόταση έτσι όπως την παρουσιάσατε. Κοιτάξτε, ε, στην Αγγλία οι φεμινίστριες ζητούν κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια. Είναι κάτι που το είχαμε, το είχαμε ζητήσει και απλώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών δεν είναι ουτοπικό αυτό που ζητάμε. Το βασικό είναι να αναγνωριστεί η συνεισφορά των γυναικών και στον επαγγελματικό τους βίο, αλλά και στην οικογενειακή του ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορέσατε να ελέγξετε τους άντρες σας. Γιατί ε, Βρετανή είναι αυτή που πήγε στο δικαστήριο και ζήτησε ίση μεταχείριση για την, για την ηλικία συνταξιοδότηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Wenn ich noch mal eine, ähm, Άλλη μία ερώτηση ας ακούσουμε. Παρακαλώ. Από την Αθήνα ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Προσπαθώ από το πρωί να καταλάβω ποια είναι η μεγάλη διαφορά αυτού του σεμιναρίου για τα θέματα της ίσης αμοιβή για ίση δουλειά από ένα σεμινάριο που θα γινόταν πριν 10 ή 15 χρόνια. Και ομολογώ ότι δεν βρίσκω τίποτα το καινούριο. Θα ήθελα να ρωτήσω η ίση αμοιβή για ίση δουλειά, αυτό το σπουδαίο σύνθημα, τι νόημα έχει κατά τη γνώμη σας σε συνθήκες παντελούς ανισότητας όταν στον ευρωπαϊκό νότο και ειδικά στην Ελλάδα η ανεργία ήδη είναι 21%, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω από τη φτώχεια προσεγγίζει το 25%, οι επικουρικές συντάξεις μέσα σε δύο μήνες μειώθηκαν κατά 50%, οι κύριες συντάξεις μειώθηκαν τρεις φορές, ε, τι νόημα έχει αυτό το σύνθημα που βάζετε ίση αμοιβή για ίση δουλειά σε ποιες συνθήκες, για ποιες χώρες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Νομίζω ότι η ερώτηση απευθύνεται σε όλα τα μέλη του πάνελ. Πρώτα η κυρία Ομινράιντον και μετά οι υπόλοιποι. Καταρχήν, σε όλες τις συνθήκες υπάρχει το άρθρο 119 το οποίο ενσωματώνει, κατοχυρώνει αυτή την αρχή. Έχουμε βεβαίως και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το άρθρο για τις ίσες ευκαιρίες και συμμεταχείριση δεν ισχύει μόνο για μισθούς και εισόδημα, αλλά και για τις συντάξεις. Θα θυμάστε ίσως ότι μάλλον το 1986 όλοι στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο κατόπιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατοχυρώσαμε την ίση αμοιβή εργασία στη χώρα μας θέμα είναι τώρα κατά πόσο κάθε φορά χρειάζεται κάποιο να προσφέρει στο δικαστήριο. Αν ζητήσετε από κάποιον ευρωβουλευτή να σα βοηθήσει, ε, βεβαίω και θα το αποκριθεί θετικά. Γιατί πολλέ φορέ η αίσθηση που έχω, φαντάζομαι και εσεί την έχετε, είναι ότι σε κάποια κράτη-μέλη ο προπολογισμό δεν είναι αυτό που έπρεπε. Δεν υπάρχει ισοσκελισμό. Και δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Από την άλλη μεριά βέβαια δεν είναι να να σηκώνουμε τα χέρια και να θεωρήσουμε ότι δεν μπορείτε εσείς να πάρετε τα ηνία των οικονομικών σας. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ μέσα σε 100%. Νομίζω ότι χέρι-χέρι θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ώστε να πάνε καλύτερα. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Πιστεύω ότι τα μέτρα που οφείλουν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη ε, με στόχο ε, να συμμορφωθούν με τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας ε, δεν πρέπει να συγχέονται με τα κριτήρια που εφαρμόζονται για να κατοχυρωθεί η ισότητα των δύο φύλων. Όπως σωστά είπατε, τι έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία. Εγώ πιστεύω πως όλοι μας ε, επιθυμούμε να είναι ταχύτερες οι αλλαγές, όλοι επιθυμούμε να είχαν συμβεί ακόμη περισσότερα πράγματα. Οι σημερινές ε, όμως ε, διαφορές δεν οφείλονται τόσο σε άμεση διακριτική μεταχείριση όσο στις νοοτροπίες που παραμένουν αμετάβλητες. Φυσικά δεν πρέπει να προσλαμβάνουμε μόνο τους νέους και τις γυναίκες και οι πιο ηλικιωμένοι ανάμεσά μας πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται. Θα πρέπει όλοι ε, να έχουν το δικαίωμα να παίρνουν γονική άδεια χωρίς να δακτυλοδεικτούνται από τους συναδέλφους τους. Αυτά είναι θέματα νοοτροπίας. Όντως όλοι θέλουμε να αλλάξουν γρήγορα οι νοοτροπίες, αλλά μήπως είναι θέμα γυρνιάς, ε, μήπως... Ε, ε, υπάρχει, πρέπει να ψάξουμε αλλού την απάντηση, γιατί από το ίδιο φίλο είμαστε και διαπιστώνω και εγώ τα ίδια προβλήματα, όπως και εσείς. Η κατάσταση ε, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Έχουμε συζητήσει επί αυτό το θέμα και χτες και σήμερα με τους Έλληνες συναδέλφους περιοριστήκαμε σε μία δήλωση αλληλεγγύης. Παραδέχομαι ότι δεν ωφελεί και πάρα πολύ μία τέτοια δήλωση. Προσπαθούμε να ε, δράσουμε επί που παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο όπως ε, της άγριας δύσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι άγρια ανατολή ε, ως προς τα ασφαλιστικά και τα συνταξιδοτικά δικαιώματα και ε, παραβιάζεται το κράτος δικαίου σε περιπτώσεις βεβαίως όπως της Ελλάδας. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε καν ποιες επιπτώσεις θα έχουν νέες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων εμείς θα θέλαμε να σταματήσει αυτή η κατηφορική πορεία και θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε και τις ε, εξελίξεις ε, στο εργατικό δίκαιο, ε, στις συλλογικέ συμβάσεις, διότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτά μίλησε η κυρία Όμιν Ρόιτεν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν και τα συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα έπρεπε ο καθένας να πρέπει να αγωνίζεται μόνος του για τα δικαιώματα του. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτό σημαντικό. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω καμία ερώτηση από το κοινό. Θα ήθελα... Να πω το εξής, σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, ε, συχνά το θέμα της ηλικία ε, συνταξιοδότησης ε, είναι ένα ζήτημα που δεν απασχολεί πολλούς μέχρι που να φτάσουν σε αυτή την ηλικία συνταξιοδότηση και ξαφνικά βρίσκονται προ εκπλήξεως όταν τελικά φτάσουν σε αυτήν την ηλικία. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αλλά σε περίπτωση που Έχουμε ένα ζευγάρι, δουλεύουν και οι δύο γονείς, ε, έχουν παιδιά και ο άντρας έχει εργαστεί περισσότερα χρόνια από τη γυναίκα, σταματάει η γυναίκα τη δουλειά για το πρώτο παιδί, στη συνέχεια μπορεί να προκύψει δεύτερο παιδί, υπάρχουν άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την φροντίδα του παιδί, ποιος θα κάτσει ε, στο σπίτι, καμιά φορά σκέφτονται ε, ε, ποιο έχει την υψηλότερη αμοιβή, εκείνος θα συνεχίσει να δουλεύει και αυτός που έχει τη χαμηλότερη θα κάτσει στο σπίτι. Συνήθως δεν είναι η γυναίκα αυτή σε φορές βλέπουμε ότι η απόφαση δεν είναι εύκολο να ληφθεί. Είναι πολλές φορές ίσως ε, όλο και περισσότερες οι περιπτώσεις που οι γυναίκες έχουν καλύτερη θέση και εκεί πραγματικά η απόφαση είναι δύσκολη. Πάντως, το θέμα της ηλικία συνταξιοδότησης σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το πιο σημαντικό, αν θέλετε, ο πιο σημαντικός παράγοντας ε, για σας, ποιος είναι. Από τη μία υπάρχουν ε, διαφορετικές σταδιοδρομίες, αν θέλετε, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε σε σχέση με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνονται στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά και το θέμα του ορίου της ηλικία συνταξιοδότησης. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, όχι? Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ποιο είναι το ζήτημα. Ε, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν όντως κάνουν διαφορετικές επιλογές ε, οι γυναίκες και οι άντρες αντίστοιχα υπό διαφορετικές συνθήκες, ας πούμε για την κατάρτιση και για την απασχόληση. Εμείς οι εργοδότες ε, θεωρούμε πως είναι θετικό να επιλέγουν οι γυναίκες σταδιοδρομίες όπως αυτή του πολιτικού μηχανικού. Εκεί χρειάζεται, χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά εργασίας, επίσης στον τομέα της ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπάρχουν κενά αλλά το δίλημα τίθεται ως εξή Θέλετε μεγαλύτερη ισότητα στην αγορά εργασίας. Αν το θέλετε, θα πρέπει οι άντρες και οι γυναίκες να κάνουν παρεμφερείς επιλογές. Αν δεν το θέλουμε αυτό, θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα συνεχίσουν να κάνουν διαφορετικές επιλογές στη ζωή τους ε, οι γυναίκες και οι άντρες και θα ε, παραμείνει και η μισθολογική διαφορά. Δηλαδή, έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας, αλλά στον επιχειρηματικό κόσμο αυτό που ζητούμε είναι όπου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση να υπάρχει και μεγαλύτερη προσφορά. Όταν όμως κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές ε, ε, οι γυναίκες σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Η περίπτωση να παντρεύεται κανείς άντρες που είναι 10 χρόνια νεότεροι και κατόπιν να κάνουν παιδιά και επειδή οι γυναίκες είναι σε καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας να σταματούν οι άντρες. Πώς σας φαίνεται αυτή η περίπτωση. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά. Έχω να σου πω το εξή. Άνοιξουμε μια ματιά στα εξοδοτικά συστήματα από πλευράς ισότητας. Νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα διαφθοράς, προβλήματα στα ταμεία. Ε, δεν είναι εδώ και ο Σνταρντέν και βλέπω, νομίζω ότι η εκπρόσωπος της Ιταλίας προέρχεται από ένα κόμμα ε, το οποίο νομίζω ότι πολλά μπορεί να μας πει για αυτή την υπόθεση. είμαι προβληματισμένος βαθιά, ενώ ότι με προβληματίζει το ποιοι εδώ μας μιλούν για τις συντάξεις. Αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι προσωπικό, δεν, είναι ερώτηση καν αυτό που σας λέω. Είναι παρατήρηση, δήλωση. Ja, Herr Dardenne hat abgesagt. Ähm, Ο κύριος Ντάρτον δυστυχώς δεν να είναι παρόν. Μας είναι πιο εύκολο να έρθουμε σε επαφή και με τους, ε, τα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου. Να δώσουμε το λόγο όμως ε, στις ομιλήτρες από το πάνελ. Κυρία Ματέρα, κοιτάξτε. Νομίζω ότι δεν κατάλαβα καλά την παρέμβασή σας, αλλά αφού μιλάμε για τα καθήκοντα των ανδρών, νομίζω ότι δεν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Θα συνεχίσω αυτά που μας έλεγε η συνάδελφος ε, από την Business Europe, ότι δηλαδή θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τις επιλογές μας ε, και να ξεκαθαρίσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Το 2011 νομίζω θα έπρεπε οι άντρες και οι γυναίκες να βρίσκονται σε θέση να κάνουν και διαφορετικές επιλογές σε σχέση με το παρελθόν. Έγινε και μια δημοσκόπηση στην Ιταλία σχετική και ρωτήθηκαν ε, πολλοί όταν γεννιέται ένα παιδί πόσο χρόνο σκοπεύει η γυναίκα να αφιερώσει στην ανατροφή πρωτού επιστρέψει στη δουλειά τη ε, και πόσο αντίστοιχα ένα ε, άντρα. Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα. Αλλά ξέρετε, ίσω θα έπρεπε όμω ε, να ασχοληθούμε με το αντίστροφο. Δηλαδή, εμεί θέλουμε την ισότητα των ευκαιριών και τον την ισότητα των, ως τα δικαιώματα. Αλλά δεν μιλάει κανείς για την ισότητα των υποχρεώσεων. Σίγουρα έχει μεγάλη σημασία και θα ήθελα να μοιραστώ αυτό μαζί σας. Δηλαδή θα δεχτούμε αυτή τη διαφορετικότητα των δύο φίλων ως προς επιλογές που κάνουν ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι όντως θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα που να μας οδηγήσουν σε περισσότερες ευκαιρίες και για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Να μπορούν να συμμετάσχουν δηλαδή από κοινού και με ισορροπημένο τρόπο και στην οικογενειακή ζωή αλλά και στην ε, επαγγελματική ζωή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει ανταγωνισμός ε, ε, οικογένεια ή δουλειά. Για τις γυναίκες αυτό το δίλημα τίθεται ακόμα θα πρέπει βεβαίως να βρεθούν λύσεις, ιδανικές λύσεις ε, ίσως δεν υπάρχουν και από κοινού θα πρέπει ένα ζευγάρι, οι δύο γονεί να αντιμετωπίσουν τη δυνατότητα αυτή ευελιξία μεταξύ οικογένειακή ζωής και επαγγελματικού τους βίου. Λοιπόν, όσον αφορά την συζήτησή μας, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να διακόψουμε, δεν έχουμε άλλη ώρα. Θα κάνουμε μία διακοπή για καφέ και κατόπιν θα μιλήσουμε για το τρίτο μας θέμα που είναι νομοθεσία που αφορά τις ε, ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών και τώρα θα διακόψουμε για μισή ώρα. <laughs> Συγγνώμη για ένα τέταρτο.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 πολύ σημαντικά που λείπουν. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Το ερώτημα είναι, χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, την ισότητα των φύλων. Έχουμε εδώ πέντε μέλη του Κοινοβουλίου, δηλαδή της νομοθετικής ε, πλευράς, αλλά και την Κάθριν Χάκιμ, η οποία πραγματικά είναι συγγραφέας ε, εξαιρετικά πρωτότυπων ε, βιβλίων το θέμα αυτό. Νομίζω ότι γνωρίζετε πια τη διαδικασία, πέντε λεπτά εισαγωγικά σχόλια και κατόπιν θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ ημών και ημών ή μεταξύ σας. Κυρία Μπάουερ, βρίσκεται αριστερά μου. Η κυρία Μπάουερ. Συγγνώμη, είναι από την Ουγγρική μειονότητα της Σλοβακίας. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Αλλά έχει γερμανικό όνομα. Ανήκει στο ΕΛΚ και νωρίτερα μα έγινε και μια παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Είστε οικονομολόγος, κοινωνιολόγος και βεβαίως έχετε εμβαθύνει σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ. Κατόπιν η Μπρίτα Τόμσεν από τη Δανία, σοσιαλδημοκράτης, που ανήκει και στην χώρα που έχει την Προεδρία. Η Δανή είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ίσης μεταχείρισης δικαιωμάτων των γυναικών. Όλες οι σκανδιναβικές χώρες είναι και θεωρούνται από πολλούς ε, το πρότυπο για τα θέματα αυτά. Η Νάντια Χίρς από την ε, Γερμανία, Ανοίξους φιλελεύθερους και είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης εδώ. Είναι ψυχολόγος και μπορεί να μας ε, παρουσιάσει κάποιες από τις πτυχές που αφορούν την ψυχολογική πλευρά αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Η Φρανσίσκα Μπράτνερ από τους Πρασίνους, Γερμανίδα. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα του, αν το επιθυμεί, το επαναλαμβάνω, από την Κοινωνική Επιτροπή. Είχαμε σήμερα το πρωί και μια άλλη συναδελφό σας από τους ε, πρασίνους που είναι γνώστης των θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες. Και έχουμε και την κυρία Τσίμερ. Η κυρία Τσίμερ επίσης είναι Γερμανίδα από την αριστερά, ειδική για θέματα απασχόλησης, κοινωνικά θέματα Και βεβαίως η Επιτροπή Απασχόλησης δεν έχει μόνο γυναίκες, αλλά ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης τα θέματα ίσης μεταχείρισης, ίσων ευκαιριών παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάτι που βεβαίως αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες. Τέλος, έχουμε και ένα μέλος του πάνελ που δεν είναι πολιτικός, είναι η Κάθριν Χάκιμ, συγγραφέας, καθηγήτρια Έχει γράψει πολλά best-seller, μοντέλα οικογενειακά της σύγχρονης κοινωνίας. Πριν από δύο χρόνια είχε έρθει εδώ και μας είχε παρουσιάσει ένα από τα βιβλία της που αφορά τα ερωτικά μοντέλα και την δύναμη στους χώρους ε, της εργασίας αλλά και στην κρεβατοκάμαρα, ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο καθένας από εσά μπορεί να μιλήσει για πέντε λεπτά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιορίσω κανένα. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο. Thank you so much. Uh, σας ε, ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να σας πω όλα αυτά που έχω κατά νου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσω. Βάσει των τελευταίων στοιχείων, προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε με διαφορά 16,4 ε, ποσοστίων μονάδων ανάμεσα στα δύο φύλλα. Δεν έχουμε πλήρη στοιχεία βεβαίως ακόμη. Από την ε, ε, στον ΝΙΑ είδαμε ότι είναι 13% και δεν έχουμε και στοιχεία από την Ελλάδα. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτές τις ε, διαφορές. Πώς ε, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας όπως, όπως τη συμφιλίωση της ε, οικογενειακής ε, και της επαγγελματικής ζωής. Τέλος πάντων, όλα αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε, αλλά το βασικό είναι να αιτιολογήσουμε αυτές τις ε, διαφορές που οφείλονται στη διακριτική μεταχείριση. Το καθήκον μας είναι να εξετάζουμε αυτές τις διαφορές στην Πολωνία έχουμε τη χαμηλότερη διαφορά, το μικρότερο χάσμα, 1,9%. Το υψηλότερο ποσοστό είναι 25,5%. και είναι το υψηλότερο ποσοστό και το ίδιο περίπου και στην, στην Αυστρία και το ίδιο περίπου στην Σλοβακία. Ποια είναι η κατάσταση επίσης όταν επιστρέφει κάποιο από την πρώτη άδεια μητρότητα. Αυξάνεται το μισθολογικό χάσμα και τιμωρείται κάποιος αντί να υποφελείται από αυτήν την ε, γονική άδεια. Πρόκειται για ένα ουσιαστικότατο κοινωνικό πρόβλημα. Βάσει της ανάλυσης μας είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ανάλογα με την ηλικία και την παιδεία παρατηρείται αυξομοίωση του χάσματος. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα σχετίζεται με την ίδια τη δουλειά ε, και την αξιολόγηση της δυσκολίας της. Ε, παραδείγματος χάρη, η ψυχολογική κόπωση των νοσοκόμων που εργάζονται στο, τμήμα, στο ογκολογικό τμήμα μιας κλινικής δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα ε, επαγγέλματα. Το είδαμε σύντομα προηγουμένως ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Θέτετε το ερώτημα αν χρειάζεται μια νομοθετική λύση. Καταρχάς θα σας απαντήσω αρνητικά. Είναι υπερρυθμισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνετε όμως όταν είναι, υπάρχει μια κείμενη νομοθεσία εδώ, η ίδια εδώ και 50 χρόνια και είναι εντελώς αναποτελεσματική. Τι κάνει κανείς. Επίσης, ε, υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα, υπάρχει οριζόντια, κάθετη, διακριτική μεταχείριση, υπάρχει το θέμα της αξιολόγησης ε, της κόπωσης, κάθε θέση απασχόλης κτλ. κτλ. Ποια είναι η δική μας ευθύνη και μπορούμε να απαντήσουμε μόνο με αυτήν την νομοθετική λύση. Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτήν την αναποτελεσματική και απερχαιωμένη νομοθεσία. Ή θα την καταργήσουμε ή θα προσπαθήσουμε να την καταστήσουμε αποτελεσματικότερη. Προσπαθούμε να προκρίνουμε τη δεύτερη λύση, να την καταστήσουμε αποτελεσματικότερη. Γι' αυτό κατέθεσα τη νέα έκθεσή μου για την ε, μισθολογική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα και εξετάζω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη νομοθεσία και δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη σε κάποια κράτη-μέλη ήπιε κυρώσει. Παραδείγματο χάρη ε, στους ε, κρατικού διαγωνισμού αποκλείονται κάποιοι όταν δεν σέβονται την νομοθεσία περί δικαιωμάτων. Το ίδιο προβλέπεται για την απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Κύρωση όταν δηλαδή παραβιάζονται οι αρχέ περί ε, των δύο φύλων. Η αγορά εργασίας ε, αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μέρες μας ε, και Από τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις περνούμε σε ένα νέο σύστημα των ε, ατομικών ή επιχειρησιακών διαπραγματεύσεων. Επίσης, τίθεται και δίδυμα ενημέρωσης. Ε, γνωρίζουμε τα πραγματικά μισθολογικά επίπεδα. Η επιχειρησιακων διαπραγματευσεων επισης ετηθηκε και διδυμα ενημερωσης γνωριζουμε τα πραγματικα μισθολογικα επιπεδα η προσβαση στη, στα πραγματικά στοιχεία νομίζω είναι αρκετά σημαντική ώστε να κλείσω έτσι την παρέμβασή μου. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την χρήση των ένδικων μέσων. Έχουμε μόνο ε, λίγες προσφυγές, ε, δηλαδή μικρή χρήση αυτών των ένδικων μέσων. Φυσικά είναι, προβλέπεται η προσφυγή, ε, η δικαστική βάση περιπτώσει η ρύθμιση των ζητημάτων, των διαφορών, ναι, αλλά αυτό συνεπάγεται και μεγάλο κόστος. Νομίζω ότι ε, μειώνοντας αυτό το κόστος θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της ε, νομοθεσίας. Και σβήνει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάουρ. Ευχαριστούμε που καταβάλλετε αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσετε όλα αυτά να μας τα πείτε μέσα σε πέντε λεπτά. Ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Συμπαθάτε με όλοι, γιατί είμαστε ε, έξι εδώ στο πάνελ και πρέπει να μειώσω αυτό το χρόνο. Έχετε λόγο. Εγώ, στα αγγλικά, θα ευχαριστήσω πρώτα απ' την κυρία Μπάουερ για αυτή την εναρκτήρια εισήγησή τη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το που μα είπε, γιατί τώρα μου έρχεται στο μυαλό η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Μα είπατε για αυτό το παράδειγμα το οποίο αφορά την συμφιλή στον συγκερασμό τη επαγγελματική με την προσωπική και κοινωνική ζωή. Κάτι το οποίο είναι πραγματικό πρόβλημα σε πολλέ χώρε και ε, υπάρχει κάτι το οποίο ισχύει. Και ισχύει και στη χώρα μου, την ε, Δανία και εκεί έχουμε χάσμα πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι Δανέζες δουλεύουν. Άλλες part-time, άλλες full-time, αλλά όλες, όλες σχεδόν είναι στην αγορά εργασίας. Ακριβώς όπως και οι άντρες. Όμως, διαφέρει πάρα πολύ το είδος της δουλειάς, διαφέρει πάρα πολύ η θέση στην ιεραρχία. Είμαστε 23η στη σχετική κατάταξη. Ακόμα και αν έχουμε πλήρη κάλυψη για ανάπηρους, για, για παιδιά, για ηλικιωμένους, Επομένως ε, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αναγκασμένες να κάνουν ε, αυτά τα πράγματα, όμως ε, ακριβώς λόγω του ότι ε, υπάρχει τέτοιο χάσμα στην αγορά εργασίας που είμαστε και εμείς θύματα αυτής της δυσμενούς παράδοσης για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία από τη Γερμανία το κληρονομήσαμε αυτό, λέω. Ξέρετε, έχω ζήσει και στην Πορτογαλία λίγα χρόνια, όπου η, χώρα, η Πορτογαλία, είναι πρώτη όσον αφορά το πόσες γυναίκες έχουν σε υψηλέ θέσει στην Και η Ισπανία είναι στο νούμερο 2 της κατάταξης. Η Δανία είναι πάρα πολύ χαμηλά και η Γερμανία είναι τελευταία όσον αφορά τη θέση αυτή. στο Max Planck, στο ίδρυμα Max Planck, ποτέ θα δείτε μια γυναίκα, α πούμε. Άλλα διαφορετικέ συνθήκε, αλλά διαφορετικοί λόγοι, γιατί οδηγούμε στο ίδιο ε, αποτέλεσμα στην κάθε κοινωνία. Αλλά θα πρέπει κανεί να το ψάξει να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο υπουργό Ισότητας κάνει δεν μπορεί ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η διχοστασία στην αγοραργασία και στην παιδεία. Να είπαμε ποιο είναι το κλειδί για να λυθεί το πρόβλημα της ίσης και της ίσης Είναι δεδομένη αυτή η αρχική και κατά το δημοτικό αλλά ακόμα δεν ε, έχουμε κάποια κριτήρια για να μπορέσουμε να να μετρήσουμε τι θα πει η ίδια αξία. Γιατί μια νοσοκόμα να παίρνει λιγότερα από έναν ε, σκουπιδιάρι ενώ έχει σπουδάσει πολύ περισσότερο. Επομένως, τελικά, όλα εξαρτώνται από το ποιος έχει καλύτερο συνδικάτο. Γυναίκε πάντω μέχρι στιγμή βγαίνουν χαμένε από οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση. Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια για τη Γερμανία, για το, το μικρόβιο που σα έχει μολύνει, το οποίο προέρχεται από τη Γερμανία. Ε, γι' αυτό και τώρα θα μιλήσουν όλο οι Γερμανίδε για να μπορέσουν να τοποθετηθούν σε αυτά που είπατε. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι αν ε, μια γυναίκα πάει στο σούπερ μάρκετ ε, σήμερα, και αγοράσει μήλα και πάει στο ταμείο και πει ότι είμαι γυναίκα και θέλω να μου δώσετε αυτά τα μήλα 20% φθηνότερα. Η απάντηση είναι τι έκπληξη θα εκφράσει ο ταμείας. Γιατί λοιπόν μία γυναίκα δέχεται να κερδίζει λιγότερο, η έκπληξή μας θα πρέπει να είναι αντίστοιχη. Ναι, χρειαζόμαστε νέα νομοθετικά κείμενα. Χρειαζόμαστε νέους νόμους γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Αλλά ο καθένας από εμά θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές και μόνο με αυτόν τον τρόπο η νόμη, η νομοθεσία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τρόπο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά από μόνοι τους οι νόμοι δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νομική βάση με το άρθρο 175 145 Και βάσει αυτού μπορεί να γίνει μια νομοθετική πρόταση που να οδηγήσει σε νέα κείμενα, σε νέα νομοθεσία. Το θέμα είναι, θα πρέπει να είναι κίνητρο ο νόμος ή θα πρέπει να εμπεριέχονται και οι κυρώσεις, οι ποινές για την μη του. Ενδεχομένως θα ξεκινήσουμε με κίνητρα όσον αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης. Έχουμε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο μια γνωμοδότηση η οποία έχει σαν σκοπό να δημιουργηθεί ένα ε, λόγο ποιότητας, μια ποιοτική αν θέλετε ε, Η ιδιότητα η οποία θα δίνεται στις ε, επιχειρήσεις αυτές που τηρούν αυτές όλες τις προδιαγραφές για τις γυναίκες. Και εγώ, παραδείγματο χάρη, πηγαίνοντας απευθυνόμενη σε μια τέτοια εταιρεία που έχει αυτό το ε, την ποιοτική σφραγίδα, είμαι κατά κάποιο τρόπο σίγουρη ότι θα τηρηθούν ε, κάποιες προδιαγραφές που με αφορούν. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα ήδη πολλά κίνητρα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να εμπλουτιστούν και να συμπληρωθούν. Αλλά για να μην ε, μιλήσουμε μόνο για την νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά αυτόν τον τομέα, θα ήθελα να πω κάτι που σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους συναδέλφους που εργάζονται εδώ σε όλες τις οδηγίες που αφορούν άλλα θέματα, άλλους τομείς, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτήν την απέτηση και αυτή την προϋπόθεση. Και πάντα θα πρέπει να αναρωτιόμαστε μέχρι πού μπορεί η συγκεκριμένη εργασία να αποκτήσει ευελιξία. Το θέμα της ευελιξίας στην εργασία είναι κάτι που πολλές φορές απασχολεί και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις γυναίκες και πολλές φορές σε διάφορες οδηγίες που αφορούν άλλα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπεριέχονται στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στις γυναίκες σε περισσότερη ευελιξία και σε καλύτερη δυνατότητα προσαρμογής. Όπως είπε και η συνάδελφος, η κυρία Μπάουερ, το θέμα των γυναικών που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από ένα παιδί, από μια εγκυμοσύνη, είναι κάτι που μας δείχνει ακριβώς το πώς έχει η κατάσταση. Οι γυναίκες σε γενικές γραμμές και κατά κανόνα βρίσκονται σε πολύ δυσχερή διαπραγματευτική θέση, για να το πούμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Φραντζέσκα Μπράτνερ. Και εγώ είμαι από τη Γερμανία. Το όσα είδαμε τα συγκρίσιμα στοιχεία από όλε τι χώρες του ΩΣΑ και είμαστε πολύ πολύ κακοί. Ίσως η Εστονία να είναι ακόμα χειρότερη από εμά, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά την ταξινόμηση των χωρών βάσει των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν από τον ΩΣΑ. Η κάθε χώρα βέβαια έχει διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές συνήθειες, και εμείς δεν έχουμε τον λεγόμενο ελάχιστο μισθό. Όλα καθορίζονται βάσει διαπραγματεύσεων και συμβάσεων σε επίπεδο κλάδου ή επιχείρησης. Αυτό βεβαίως δίνει μεγάλη ευελιξία. Εγώ σήμερα άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από τους προηγούμενους ομιλητές και όσον αφορά την κοινή μισθοδοσία όσον αφορά τους ίσους μισθούς και τις διαφορές που σήμερα υπάρχουν, που φτάνουν μέχρι και το 50%, βλέπουμε ότι όλες οι πολιτικές ε, ομάδες, από τους πράσινους μέχρι τους κέντροδεξιούς, στηρίζουν την βασική αρχή που διεκδικούν και ζητούν οι γυναίκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που υπάρχει στη συνθήκη του Άμστερνταμ, που είναι ίση αμοιβή για ίση εργασία. Αυτό είναι κάτι που στην πράξη βεβαίως βλέπουμε ότι απέχει πάρα πολύ από τα κείμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό που ζητάμε εμείς σήμερα είναι να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν οι διάφορες μισοδοτικές κατηγορίες, το ξέρουμε αυτό, η σύγκριση των στοιχείων θα πρέπει να είναι εφικτή, άρα περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όπου σήμερα υπάρχει ακόμα μία δυσχέρεια στο ανακοινωθούν οι μισθοί και οι αμοιβέ των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε σε πολλές χώρες, όχι μόνο στη Γερμανία. Και μπορεί να βελτιωθεί το θέμα της διαφάνειας. Και βεβαίως Στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, έχουμε στοιχεία που δείχνουν την δυσκολότερη κατάσταση των γυναικών ανάλογα με το σε ποια κατηγορία ανήκουν, ανάλογα με το αν ε, είναι μετανάστες ή όχι. Και επαναλαμβάνω ότι αν είχαμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερα στοιχεία θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την κατάσταση μεταξύ των επιχειρήσεων, μεσαίων ή μεγάλων. Και θα βλέπαμε ότι πολλές φορές πολλά εξαρτώνται και από την δίκηση των επιχειρήσεων. Δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι προσφυγές δεν υπάρχουν ε, γυναίκες που προσφεύγουν σήμερα και πολλές φορές η αντιμετώπιση αν θέλετε, προς μια γυναίκα η οποία θα αποφασίσει να προσφύγει γιατί ο μισθός της είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ενός άντρα, είναι κάτι που πάρα πολύ σπάνια το βλέπουμε. Καμία γυναίκα δεν θέλει να την στιγματίσουν. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες συλλογικές ε, προσφυγές. Μία ομάδα γυναικών, αυτό βεβαίως συμβαίνει συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο ίσως έχει και περισσότερη βαρύτητα μια τέτοια προσφυγή. Τρίτο σημείο, οι κυρώσεις. Βλέπουμε επίσης ότι σε περιπτώσεις προσφυγών οι κυρώσεις, αν θέλετε, που επιβάλλονται στους εργοδότες είναι πολλές φορές χαμηλότερα ποσά από την εξοικονόμηση που κάνουν μη πληρώνοντας ε, ίδιους μισθούς τους άνδρες και τις γυναίκες. Και εδώ όμως υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τη μια χώρα στην άλλη. Θεωρούμε και εμείς ότι αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπράτνερ. Και συνεχίζουμε ακόμα πιο αριστερά. Κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ. συνεχίσω τώρα. Εγώ κοίταξα το πρόγραμμα και είδα ότι ακούσαμε αναλύσεις, στοιχεία, αριθμούς. Εγώ μπορώ να συνεχίσω την παρουσίαση του θέματος αυτού αναφερόμενη σε μια γνωμοδότηση την οποία επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της έκθεσης που προετοιμάζει η Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο πτυχές αυτού του θέματος. Κάτι που αφορά το θέμα των δεσμευτικών ή μη δεσμευτικών μέτρων. Το χάσμα μεταξύ των αποδοχών των μισθών θα γεφυρωθεί εάν και εφόσον μπορέσουν οι γυναίκες να αλλάξουν τη θέση τους στην κοινωνία. Το θέμα της διαφορετικής μισθοδοξίας δεν εξαρτάται βεβαίως μόνο από την ιεραρχία στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, αλλά και από το τι πρόσβαση έχουν οι γυναίκες, τι δυνατότητες, τι δικαιώματα έχουν οι γυναίκες γενικότερα σε μια κοινωνία, άρα και στην αγορά εργασίας και πόσο σοβαρά τις λαμβάνουν υπόψη τους. Γιατί παραδείγματος χάρη σήμερα βλέπουμε ότι οι γυναίκες κάνουν καλύτερες σπουδές, το 75% των ε, γυναικών που βγαίνουν από ανώτατα ιδρύματα, πανεπιστήμια, ανώτατες ε, σχολές, συνεχίζουν να λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές από τους αντίστοιχους άντρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης μόρφωσης των γυναικών, αντίθετα mm. δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την ε, μισθοδοσία και τη θέση τους μέσα στις επιχειρήσεις. Από την άλλη μεριά, διαπιστώνουμε επίσης ότι σε διάφορα επαγγέλματα είναι παντελώς απούσες οι γυναίκες. Και αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε ελλειπή κατάρτιση, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα. Από τη μία μεριά λοιπόν βλέπουμε ότι οι γυναίκες με ίσες δεξιότητες, προσόντα και διπλώματα ανώτατης εκπαίδευσης δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν μια οικονομική ανεξαρτησία και από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές να συγκεράσουν και να αντιμετωπίσουν από κοινού και με ικανοποιητικό τρόπο την οικογενειακή τους και προσωπική τους ζωή με μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει μια αλλαγή στην αντιμετώπιση των γυναικών από την κοινωνία αν δεν υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές καινοτομίες, καινοτομίες στην αγορά εργασίας, πρόοδη σημαντική, που να αφορούν τις γυναίκες, αποκλειστικά τις γυναίκες, που να τις επιτρέψουν να προχωρήσουν. Και βλέπουμε σήμερα ότι με την λιτότητα, με την οικονομική κρίση, τα θέματα αυτά είναι λιγότερο στο προσκήνιο. Και ότι οι επιχειρήσεις έχουν άλλα προβλήματα και δεν πρόκειται εθελοντικά και από μόνοι τους να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και σας ζητώ το Κοινοβούλιο να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιπτώσεις σε χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση όπως η Ισπανία και η Ελλάδα ποιες είναι οι επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας και της οικονομικής κρίσης επί των γυναικών, οι οποίες εργάζονται με αντίξωες συνθήκες, με αβεβαιότητα και πώς εξελίσσεται η επαγγελματική ζωή των γυναικών σε αυτές τις συνθήκες μέχρι την συνταξιοδότησή τους. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ουσιαστική συζήτηση πολύ πιο ουσιαστική από το αν χρειάζονται ναι ή όχι περισσότερα νομοθετικά κείμενα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσίμερ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, εσείς ε, μας παρουσιάσατε το θέμα από μια καθαρά κοινωνική πτυχή. Και θα δώσω το λόγο στην Κάθριν Χάκιμ, η οποία δεν είναι πολιτικός, όπως είπα και προηγουμένως, και είναι συγγραφέας. Έχετε πέντε λεπτά. Ασχολούμαι με τα θέματα των γυναικών και συγκεκριμένα τα, τα εργασιακά θέματα και τα τομιστορικά χάσματα, όλα αυτά, όλη η θέση στην όλη μου τη ζωή, όλη μου την επαγγελματική διαδρομή, όλα αυτά τα έκανα και αυτά τα οποία εγώ θέλω να σας πω περιέχονται σε αυτή την έκθεση που έχω συγγράψει για το κέντρο μελετών, υπάρχουν στο σχετικό website και επίσης υπάρχουν ε, και στο κέντρο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου έδωσε ένα αντίτυπο. Ποιο είναι το, το, το ζουμί, ότι μπορεί να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτό το μισθολογικό χάσμα. Το ζήτημα είναι ότι μόνο το, το μισό εξηγούν και, και το μισό μόνο που είναι μια δυσμενής διάκριση. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα Οπότε τότε μπορούμε να εξηγήσουμε το σύνολο αυτού του, του, αυτού, του προβλήματος. Δηλαδή έχουμε κάποια, κάποια στοιχεία τα οποία έχει στα, στα χέρια της Κομισιόν υποχρεωμένα να τα χρησιμοποιήσει γιατί είναι υποχρεωμένη να υπολογίσει, δεν βοηθούν καθόλου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι, το αντίθετο είναι παραπλανητικά. Επίσης θέλω να σας πω πως ε, ε, τώρα επιβάλλει κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικά και τα οποία αυτά είναι αποτελεσματικά εάν, εάν όμως ε, εφαρμοστούν γιατί σε πάρα πολλές χώρες αυτά παραμένουν νεκρό γράμμα. Δεν υπάρχει εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας για με αυτά και ένας λόγος για τον οποίο έχουμε αποτελέσματα στην Βρετανία είναι διότι εδώ εμείς στη Βρετανία ε, έχουμε δικαστήρια όπου μπορούν να πάνε γυναίκες μαύροι ε, να, να, να, καταγγείλουν τη, δυσμενή διάκριση από τη βάση του φίλου, του, επί τη βάση της θρησκείας οτιδήποτε. Και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κανείς να πληρώσει μία δεκάρα, μία πένα. Βέβαια. Έχει και αυτό το σύστημα της ε, ε, δωρεάν δικαιοσύνης, όμως ε, αυτό τους, τους ταρακουνάει τους εργοδότες, γιατί έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να επικαλεστούν τέλο πάντων με το τη σχετική νομοθεσία. Αν επομένω υπάρχει σύστημα ουσιαστική εφαρμογή, ε, τότε βοηθάει ο νόμο, τότε έχουμε αποτελέσματα, οπότε στην Βρετανία έχουμε δει τέτοια αποτελέσματα και έτσι μπορείτε να διαπιστώσετε τι γίνεται με αυτό το μισθολογικό χάσμα και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα θεσμού διάκριση. Ε, ε, εγώ έχω δει περιπτώσει κατά τι οποίε όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διακρίσεις, ας πούμε φαρμακεία, μετάφραση και μιλούμε για κάποια ε, επαγγέλματα τα οποία είναι συνήθως ε, απασχολούν ευρύτερο κόσμο από ότι ο εθνικός μέσος όρος. Επομένως, ε, το θέμα είναι το είδος της δουλειάς, το αν κανεί δουλεύει part-time ή όχι. Πρόκειται όμω για κάποιε πραγματικέ ουσιαστικέ επιλογέ που θα πρέπει να κάνει κάποια γυναίκα και πρέπει κανεί να σεβαστεί αυτέ τι επιλογέ. πάρει κανεί να σταματά και να λέει ε, θα πρέπει να, το δούμε σαν συνδυσιακό θέμα, θα πρέπει κάποιο να, να, να συνειδητοποιηθεί. Τέλο πάντων, θα έχω εξετάσει όλα, όλα όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών ε, και επίση ε, έχω και ένα άλλο βιβλίο για τη θεωρία την μισιακή Έχω κάτσει και έχω εξετάσει όλες τις χώρες της ε, ΕΟΚ, ε, του ΟΣΑ και το τι γίνεται στα κράτη της Βορείου Αμερικής και συνολικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφοροποιημένες ε, συμπεριφορές, αξίες, στόχοι. Υπάρχει μία μειονότητα γυναικών που θέλουν σταδιοδρομία. Ε, ο ακριβώς όπω τη θέλουν κυνηγάνε, είναι φιλόδοξες όπως και οι άντρε έχουν κίνητρο και φτάνουν πάρα πολύ ψηλά, όμως είναι μόνο το 20% όσον αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στη Σουηδία, ακόμα και αν ή στην Σουηδία έχουμε περίπου 30% των γυναικών οι οποίες δουλεύουν full time συνέχεια σε όλους τις με ζωή. Και αυτό είναι με την καλύτερη νομοθεσία παγκοσμίω που έχει η Σουηδία. αφού δεν, δεν υπάρχει το κέντρο στη Σουηδία, δεν μπορεί να υπάρξει πουθενά. Η παιδεία, επομένω, δεν είναι η λύση. Γιατί τώρα οι, οι γυναίκε έχουν καλύτερη παιδεία από του άντρε. Και συνεχώ διαλέγουν τα λάθο μαθήματα, τη λάθο σχολή. Δεν πάνε να γίνουν ούτε μηχανικοί, Ούτε λογιστές, ούτε δικηγόροι όπως οι άλλοι, διαλέγουν τη φιλολογία, γλώσσες, ιστορία της τέχνης και όλα αυτά τα, τα, τα, τα, μαθήματα της επιστήμης που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αλλά που δεν έχουν την ίδια εμπορική αξία. Να γιατί ούτε η παιδεία πρόκειται να κάνει την διαφορά. Ούτε κάνει, ούτε θα κάνει. Επομένω, εγώ στο βιβλίο μου αναπτύσσω το επιχείρημα ότι οι ευκαιρίε δεν πρόκειται να μα ε, δώσουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα, διότι τώρα συνεχώ μιλούμε για το τι θα γίνει με αυτό το, το χάσμα το μισθολογικό και λέμε για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κάποια ε, δίκαια μέτρα. Όχι, δεν, δεν μας βοηθά αυτός ο συλλογισμός. Ίσες ευκαιρίε είναι άλλο πράγμα και ίσα αποτελέσματα είναι άλλο. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να αποσπάσετε αποτελέσματα ισότητα εάν κάποιο δεν έχει ουσιαστικές επιλογές, ουσιαστικά εναλλακτικά σενάρια. Είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα. Ένα από αυτά τα οποία εγώ εξηγώ στην έρευνα που έκανα είναι ότι στι χώρε που έχουν λιγότερη ισότητα μεταξύ των δύο γυναικών, όπως ας πούμε τις αγγλοσαξονικές χώρες, η Αγγλία, τότε οι γυναίκες ε, είναι πιο πιθανό να φτάσουν στο, ε, στις υψηλότερες θέσεις της ε, ιεραρχίας. Περισσότερο παρά στις χώρες που έχουν φανταστικές πολιτικές ισότητας όπως η Σκανδιναβία. Και αυτό είναι γεγονός. Αυτό το, το, το, το απέδειξα. ότι η Σκανδιναβία και, η Σκανδιναβία και άλλοι, και άλλοι μελετητές το έχουν αποδείξει. Δεν υπάρχει εμβολία. Επομένως, οι πολιτικέ ισότητα των φύλων δεν πρόκειται να αποδώσουν, να μα οδηγήσουν αντίστοιχα αποτελέσματα, ούτε πρόκειται να συρρυκνώσουν αυτό το πιστολογικό χάσμα. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να τα ξανασκεφτούμε. Είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τι γυναίκε για να πετύχουν περισσότερα και να πάρουν καλύτερε θέσει στην, στην, στην αγορά. Ε, και με τι πολιτικέ Είναι πολιτικέ οι οποίες ε, αποδίδουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ρύθμιση σε ενωσιακό επίπεδο. Και όμως αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε σε ενωσιακό επίπεδο είναι να δούμε πώς όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν κάποια νομικά συστήματα τα οποία να επιβάλλουν ε, τις υπάρχουσες ίσες ευκαιρίες, να εφαρμόζονται οι νόμοι κατά των δυσμενών διακρίσεων και αν αυτό γίνει τότε θα έχουν πλατεσμάτα. Θα μπορούσα να σας πω επίσης τι είδους πολιτικές θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες, περισσότερα αποτελέσματα για την κατάσταση των γυναικών στην αγορά απασχόληση, αλλά πάντα μιλάμε σε εθνικό επίπεδο και δεν συζητούμε αυτό τώρα. Συζητούμε τι πολιτικέ τη Ενωσιακή. Άρα εδώ βάζω τελεία. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ε, είναι, ήταν κάπως προκλητικά τα σχόλια σας, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι ε, θα ακούσουμε περισσότερες ερωτήσεις. Ε, σε σχέση ε, με την ε, αυτοανάλυση που πρέπει να κάνουν κάποιοι επιτόπου στα κράτη-μέλη, όπω τη χώρα μου παραδείγματο χάρη, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να δώσω τη δυνατότητα στου μετέχοντες να θέσουν ερωτήσει. Έχετε έξι μέλη ε, στο πάνελ, εξέδεσαν τι απόψει του. Μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα σα. Υπάρχει διερμηνία. Μπορείτε να μιλήσετε διάφορες γλώσσες αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά. Παρακαλώ. Να συστηθείτε σας παρακαλώ πριν την ερώτηση. Είμαι δημοσιογράφος από την Γερμανία, το όνομα μου είναι Ντούρν. Μιλήσατε για την άνηση αμοιβή για αντίστοιχες εργασίες. Εγώ ξέρω όμως ότι στη Γερμανία υπάρχουν ε, στοιχεία από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν κάνει κάποιες μελέτες και δείχνουν ότι παραδείγματος αν για μηχανικούς οι αμοιβέ δεν είναι διαφορετικές για ίση εργασία. Τι έχετε να πείτε. Κοιτάξτε, η απάντηση μπορεί να είναι πολύ απλή και σύντομη. Αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι, μπορεί. Νομίζω ότι πρόκειται για αμυγός διακριτική μεταχείριση στις βόρειες χώρες, στη Δανία, στη Γερμανία. Υπάρχουν ε, λιγότερες γυναίκες μηχανικοί από ότι άντρες. Στη Νορβηγία, όπου είναι πολύ προχωρημένη ως προς την νομοθεσία για την καταχείριση των δύο φύλων, έχουν θεσπίσει ένα σύστημα βάσει του οποίου κάνουν την αξιολόγηση. Δεν λέω ότι ο μηχανικός πρέπει να πληρώνεται καλύτερα από ε, το, την τον υπεύθυνο ενό ευρωφωνηπιακού σταθμού. Υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται, μα έχω σπουδάσει περισσότερα χρόνια, γιατί ε, ε, είναι χαμηλότερος ο μισθός μου. τελικά, σε μια σχετική προσφυγή κέρδισε η ενάγουσα την υπόθεση και το αναφέρω αυτό διότι τίθεται ζήτημα αξιολόγησης ε, των διαφόρων θέσεων εργασίας. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε. Θα έλεγα, λέει η κυρία Χάκιν, ότι εξαρτάται από το πώς λειτουργεί και το δικαστήριο. Δηλαδή, χρειαζόμαστε ένδικα μέσα. Χρειάζεται να υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσφυγής ε, και δεν προβλέπεται αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ε, τα ειρηνοδικεία θα πρέπει να ε, λειτουργούν με απλό τρόπο, να είναι εύκολο για τους πολίτες. Να προσθέσω κι εγώ ότι όλα καλά είναι αυτά που λέμε και ωραία, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι Εντάξει να υπάρχουν τα ένδικα μέσα, αλλά θα χρησιμοποιούνται. Πώς θα χρησιμοποιούνται, θα είναι ευχερές για τους πολίτες. Ε, στην ε, Γερμανία έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, ανακλάδο και φυσικά τα συνδικάτα φροντίζουν να είναι ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά και η... δεν, μπορεί, δεν μπορεί δηλαδή να παρέμβει το κράτος μέσω της νομοθετικής οδού. Είναι όλα αποφασίζονται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις από τους εργοδότες και τα συνδικάτα των εργαζομένων. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, τρόποι για να αντιδράσουν οι πολίτες της κάθε χώρας ε, και νομίζω ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν συλλογικές αγωγές, όχι μεμονωμένες. Ε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε βεβαίω ότι κατοχυρώνεται η ισότητα μόνο και μόνο επειδή είναι συλλογικέ οι διαπραγματεύσει. Υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις, όπως είπαμε, η αμοιβή κάθε δουλειά. Ε, Είπαν κάποιοι ότι επιλέγουν οι γυναίκες σε πιο θέσεις εργασίας με χαμηλότερες ε, αποδοχές σε σχέση με τις ε, σταδιοδρομίες ε, που επιλέγουν οι άντρες. Μήπως πρέπει να έχουμε μια ρήξη με το παρελθόν και να αλλάξει αυτό το πρότυπο. Ναι, αυτό το θέμα συζητήθηκε και στο πρώτο πάνελ. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία αμείβονται καλά και στα οποία δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες. Ή όταν ξαφνικά πολλές γυναίκες ε, προσχωρήσουν στο επάγγελμα αυτό, ξαφνικά μειώνεται η αμοιβή. Γίνεται ένα υποβαθμισμένο επάγγελμα. Προέρχομαι από την Ουγγαρία, είμαι δημοσιογράφος και έχω την εξή ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, μετά από κάποιο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν πολιτικοί που μπορούσε να ασκήσει κανείς. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο στο τι μπορούμε να πετύχουμε κάποια πολιτική. Και κατόπιν θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι ορισμένα πράγματα απλώς δεν γίνονται με πολιτικές. Εάν σας κατάλαβα καλά, επαναλαμβάνω, έχετε μια λίστα από τις αναγκαίες πολιτικές, τι θα μπορούσε να κάνει κάποια χώρα τι πολιτικές μπορεί να χαράξει μια χώρα και τα υπόλοιπα να τα αφήσει στην αγορά. Α, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Οι υπάρχουσες πολιτικές είναι το ελάχιστο. Ο ελάχιστος μισθός και ελάχιστη αμοιβή όπου θεσπίστηκαν είχαν επιπτώσεις στο πόσα κερδίζουν οι γυναίκες. Γιατί είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες παρά οι άντρες στην ζώνη των, των ελαχίστων αμοιβών. Ίσως ευκαιρίες απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης, όλες αυτές είναι βασικές ε, νομοθεσίες, και αναγκαίες. Υπάρχουν αυτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό επευλήθη. Και κατά κάποιο τρόπο και σε εμά επευλήθη όπως και σε άλλες χώρες. Και όλες οι χώρες δυσκολεύτηκαν βέβαια να ε, τα αποδεχτούν, αλλά φυσικά θα πρέπει όλα να εφαρμοστούν και πρόκειται για κάτι το οποίο συστηματικά το παραβλέπουμε. Δηλαδή, πόσοι επιφορμοί σε κάθε χώρα. Υπάρχουν ε, εργατοδικεία, είναι φτηνή προσφυγή εκεί, ε, ομαδικές αγωγές, συμφωνώ. Καμιά φορά βοηθούν. Πολλέ φορέ ε, δεν θέλει κάποιο να εκτεθεί ασχόντα αγωγή, αλλά έτσι αισθάνονται καλυμμένοι από την ομάδα. Είναι θέμα δικονομία επίση. Επομένω, πολλέ φορέ ενθαρρύνεται έτσι μια επιθετική στάση για την επίλυση προβλημάτων. Ο ένα θα έλεγε ότι δεν πρέπει κανεί να τσακώνεται, υπάρχουν καλύτεροι τρόποι. Συμφωνώ. Η ανατολίτικη προσέγγιση η πειθός, η συζήτηση, η προσπάθεια εξέβρεση συνένεσης είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερη προσέγγιση, πιο πολιτισμένη. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ίσως είναι καλύτερο. Και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πολιτική πάντως από πλευρά, της συμφιλίωσης της οικογενειακής και της οικογενειακής ζωής νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει σε αυτό το επίπεδο εθνική πολιτική. Ένα παράδειγμα το, το, το, πώς λειτουργούν τα σχολεία. Ο χρόνος. Η κάθε χώρα έχει το δικό της πρόγραμμα. Και ποτέ δεν βοηθάει αυτό τους γονείς. Την Τετάρτη απόγευμα στη Γαλλία πάνε πίσω, τα παιδιά νωρί, στην Αγγλία το, το μισό, τη μισή εβδομάδα γυρίζουν το απόγευμα σπίτι, στη Γερμανία πρέπει να γυρίσουν για γεύμα και μετά να ξαναπάνε σχολείο μπλοκάρεται τη μαμά και το ίδιο και για τις σχολικές διακοπές. Ε, η προέλευση είναι με μια γεωργική κοινωνία που προβλέπει. Θα πρέπει να είναι μικρότερε διακοπέ και πιο συχνά και, και προστατευμένε προ Πάσχα και Χριστούγεννα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα που μπορούν να τα ρυθμίσουν οι εθνικέ κυβερνήσει και θα κάνουν τη διαφορά. Και, και, και, όχι μόνο για τι μανάδε, και μάλιστα για του πατεράδε. Δεν είναι αυτά θέματα για κοινωνική νομοθεσία. Όμω από την άλλη μεριά ε, θα έχουν πάρα πολύ σημαντικέ. επιπτώσει. Ξέρω ότι το θέμα αυτό ε, διχάζει, υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά όπου τυχόν υπάρχουν και τέτοιες ρυθμίσεις, ας πούμε στι κάτω χώρε. Ε, το να δουλεύει κανένα part-time χωρί χωρίς να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Και στο Βέλγιο Επίση υπάρχει μια πολιτική που θεσπίσανε όπου οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει να δουλεύει part-time για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς να επικαλεστεί κάποιο λόγο. Άρα δεν θα έπρεπε ούτε άντρε ούτε γυναίκε να βρουν κάποια δικαιολογία. σε αυτό το χρησιμοποιούν και άντρε και γυναίκε και έτσι αλλάζουν οι νοοτροπίε και το πώ συμπεριφέρεται ο κόσμο. Ήρεμα, ομαλά, βαθμιαία, χωρί να υπάρχει συγκρουσιακή προσέγγιση ούτε και δίκες και δικαστήρια much. I don't right now, please. If you have a question, please raise your hand up clearly. Αν έχετε ερώτηση, σηκώστε το χέρι σα. Αλλά ξεκάθαρα, μην, μην, μην, μην ε, τυχόν τεντώνεστε και νομίζουμε ότι σηκώστε το χέρι. Έχετε το λόγο. Προς εσάς απευθύνεται η ερώτησή μου, κυρία Τσίμερ. Είπατε ότι δεν αρκούν ε, οι νομοθεσίες, τα διατάγματα, οι κανονισμοί και θα πρέπει οι ίδιες οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν διαφορετικά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά ακούσαμε πολύ καλά ότι χωρίς την απαραίτητη νομοθεσία που να πλαισιώνει τη θέση των γυναικών, οι γυναίκες είναι αυτές που τελικά θα χάσουν, θα είναι οι χαμένες ε, αυτής της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Επανειλημμένα με έχουν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι ποιες είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για τις γυναίκες. Σίγουρα πλήσει τις γυναίκες περισσότερο τους άντρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, στην Αγγλία περισσότερο πλήσονται οι άντρε παρά οι γυναίκε. Και από ό,τι κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε κάποια μελέτη και παραδέχεται ότι περισσότερο πλήσονται οι άντρες περισσότερο από τις γυναίκες κατά μέσο όρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στερεότυπο ότι πάντοτε θύματα είναι οι γυναίκες. Όχι. Οι άντρες πλήσονται περισσότερο, υποφέρουν περισσότερο σε όλες τις κρίσεις. Συνήθως έχουν στις περισσότερες χώρες γυναίκες και παιδιά να θρέψουν. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι το να χάσει τη δουλειά τη μια γυναίκα α, ψυχολογικά την, την θίγει λιγότερο από ότι τον άντρα. Πάντως, τέλο πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι η ύφεση έχει πλήξει περισσότερο τους άντρες. Ähm, το θέμα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ε, η νομοθετική ρύθμιση δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις και να καλύψει όλα τα κενά, να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα μείγμα από νομοθετική ε, ρύθμιση και από μέτρα που να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις γυναίκες να δουν διαφορετικά την ε, κατάστασή τους. Ένα ερωτηματολόγιο στην Όπελ έδειξε ότι οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες εργαζόταν εκεί ήταν είτε με μερική σύμβαση εργασίας είτε σε σχέση υπεργολαβίας με την εταιρεία και μάλιστα οι ε, χαρακτηριστική απάντηση των γυναικών είναι ότι επιθυμώ αυτόν τον τύπο εργασίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι οι γυναίκες που επιθυμούν να εργάζονται με μερική απασχόληση θα πρέπει να είναι συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να βασίζονται σε συμβάσεις εργασίας με την απαραίτητη εγγύηση και τις ε, προδιαγραφές που επιθυμούμε και για ένα κανονικό επάγγελμα με πλήρη απασχόληση. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ε, αν χρειαζόμαστε ναι ή όχι ένα, μια ποσόστοση για τις γυναίκες. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, όταν προσπαθούμε να μετρήσουμε την ε, αντιμετώπιση των γυναικών βλέπουμε πολύ αντιφατικά αποτελέσματα. Το θέμα των ποσοστώσεων είναι κάτι που θα πρέπει πραγματικά να ρυθμιστεί με ένα μείγμα νομοθεσίας, μέτρων, κινήτρων. Για μένα δεν είναι σημαντικό αν χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά αν τα νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν και εφαρμόζονται είναι κατάλληλα και προσφέρουν τις απαραίτητες εγγύησεις στις γυναίκες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Μπάουερ και κυρία Τόμψεν. θα σας πω ότι δεν μπορούμε όλα να τα νομοθετήσουμε. Στη χώρα μας πιστεύουμε ότι οι άντρες και γυναίκες είναι ίσοι και έχουμε διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι όταν κάποιος άντρας πάει κάπου που κυρίως δουλεύουν οι γυναίκες, όμως, ας πούμε πάει να γίνει νοσοκόμος, θα γίνει επικεφαλής μέσα σε δύο μήνες. Το ίδιο γίνεται και στους παιδικούς σταθμούς. Περισσότερο μετράνε οι άντρες. Να, και, στα συνδικάτα στη Δανία. Το ίδιο γίνεται. η αρχηγοί των συνδικάτων είναι οι άντρες. 80% του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άντρε. Οι ίδιες οι γυναίκε ψηφίζουν τους άντρε και θεωρούν λοιπόν τελικά ότι μετράνε περισσότερο από αυτέ. Αν πάει μια γυναίκα να δουλέψει σε ένα συνεργείο, α πούμε, που θα, στον, πά, πάτο θα, θα της θα βρεθεί και θα μείνει. Ήδη αυτά από την παιδική ηλικία φαίνονται. Τα δεκάχρονα αγοράκια παίρνουν διπλάσιο χαρτζηλίκι από τα κοριτσάκια. Άρα πρώτα πρώτα θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να συνειδητοποιηθούν οι γυναίκε. οι, μα, μαμάδες τι κάνουν με τα παιδάκια τους. Χωριστά παίζουν τα αγοράκια, χωριστά τα κοριτσάκια και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Για αν θέλουμε την πραγματική ισότητα. Δεν είναι δυνατόν η ισότητα να οφείλεται μόνο στην ε, νομοθεσία. Yes. <clears throat> Thank you very much. I... Και πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα απευθυνθώ στην κυρία Μπάου για ένα από αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα που είπε και η κυρία Τόμσεν. Για πέστε μας. Πώς θα μετρήσουμε, πώς θα αποτιμήσουμε την εργασία, πώς θα αξιολογήσουμε την εργασία. Άκουσα μέσα όλα παραδείγματα. Αν λοιπόν κάνουν ακριβώ την ίδια δουλειά οι γυναίκε, από ό,τι φαίνεται πληρώνονται διαφορετικά. Να, το, το μισθολογικό χάσμα. Αν όμω έχουμε δύο διαφορετικέ δουλειέ, μία να είναι νηπιαγωγό και κάποιο να είναι μηχανικό σε συνεργείο. Πώ θα μετρήσετε πόσο μετράει, πόσο αξίζει κάθε δουλειά. Για πετε μα και εσεί που έχετε την έκθεση τη σχετική, Πώ θα μετράτε αυτά. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Και ε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έχουμε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο αφορά την ε, περίοδο επόμενη ε, γιατί είναι τελικά μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση όλα αυτά να τα αξιολογούμε γιατί όντως Όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει είναι κάποιες διαφορές που είναι δικαιολόγητες. Υπάρχουν κάποια σωματικά χαρακτηριστικά όπως η σωματική δύναμη και άλλες ε, δεξιότητες και ιδιότητες υποτιμώνται. Ας πούμε, η υπευθυνότητα για τους ή τις ταμείες. Εγώ θέλω να πω το εξή για την κουβέντα μας. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μας δίνει το ελάχιστο στάνταρ, το μήνυμα, τον ελάχιστο, την ελάχιστη ρύθμιση. Για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ εύστοχο το παράδειγμα που είπαμε για το Ηνωμένο Βασίλειο για την ελεύθερη πρόσβαση την, τη δωρεάν προσφυγή στη δικαιοσύνη και έτσι δεν υπάρχουν δυσμένες διακρίσεις από πλευράς πληρωμής. μπορεί να υποχρεώσουμε κανένα κράτο να κάνει το ίδιο. Όμω μπορούμε να του πούμε ότι θα πρέπει η πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη να γίνει ευκολότερη. Και έτσι θα πρέπει να μπορούν οι αρχές να εξετάζουν κάθε φορά πώς εφαρμόζεται αυτή η αρχή που καταχρώνεται στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε μια συνταγή λεπτομέρειε στο τι πρέπει να κάνει κάθε κράτο μέλο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε, να βρούμε τα, τα ελάχιστα στάνταρ, του ελάχιστου κανόνε για το πώ μπορούν όλα αυτά να τα ρυθμίσουν. Γιατί ε, αυτό θα, θα μας οδηγήσει έτσι σε αδιέξοδο. Αλλού χρειάζεται νομοθεσία, άλλου δεν χρειάζεται. Όντω από το 1957 υπάρχουν νόμικοι και διατάξεις και δεν έγινε και τίποτα. Η πρόεδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φραντσέσκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ονομάζομαι Κατελίνα Καρμόνα και είμαι από την Βαρκελόνη, την Ισπανία και θα ήθελα να σας ε, πω το εξής διαπίστωσα ότι σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία το κράτος προνοίας συρρυκνώνεται και η προσβασιμότητα επίσης σε παιδεία και υγεία και φροντίδα των ανηλίκων τελικά όλα αυτά πάνε και μετακυλούνται στις γυναίκες. Γι' αυτό και προβληματίζομαι. Για πέστε μας, τι θα γίνει με αυτή την ε, πρόκληση, πώς μπορεί να βρούμε μια λύση σε αυτή την κατάσταση, πώς, πώς, πώς μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Η ερώτηση αφορά όλους το πανέλ, δεν είναι. Ωραία. Εξ αριστερών. Νάντια. Κοιτάξτε. Αυτά είναι γνωστά φαινόμενα. Στη Γερμανία, ας πούμε, ήταν αυτονόητο ότι θα κάνουν τον οικοκυριό και θα μεγαλώνουν τα παιδιά γυναίκες. Σήμερα, όμως, δεν γίνεται έτσι. Έχουν συνειδητοποιήσει οι άντρε πόσο αξίζει η δουλειά στο, στο σπίτι των οικοκυριών. Ας πούμε τώρα, χρησιμοποιούν περισσότερο το καθαριστήριο, τι καθαρίστριε κλπ. Οπότε τώρα έχει, να, πώς αποτιμάται η δουλειά στο νοικοκυριό. Επομένως βλέπετε τι γίνεται. Όντω υπάρχει συρρήγνωση του κράτου προνοίας, όπως είπατε. Το ερώτημα είναι αν οι γυναίκες θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία επειδή παραδείγματος χάρη κλείνει ένα νηπιαγωγείο, ένας βρεθικός σταθμός, τι θα κάνουν από εκεί και πέρα, πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει ή δεν υπάρχει έτσι ώστε να τοποθετηθούν στην κοινωνία από τη που θα χάσουν την παροχή μιας υπηρεσίας. Και αντίθετα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάθε γυναίκα πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό της προς τα ποια κατεύθυνση θέλει να πάει. Αν θέλει να ασχοληθεί με τα παιδιά της, αν θέλει να τα αναθέσει στους γονείς της ή σε κάποιον άλλο φορέα ή κάποιον άλλο άνθρωπο. Είναι κάτι που σαφώς έχει επιπτώσεις ε, και σε άλλα επίπεδα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι οι περικοπέ του κράτου προνοία πρόκειται να έχουν επιπτώσει ε, στην κατάσταση των γυναικών. Αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι στη Δανία ε, τέλη δεκαετίας του 60 θα πρέπει να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας γι' αυτό διότι προσέφερε την κάλυψη των παιδιών το, το, το, το, το, κράτος 100% κάλυψε δεν ήταν υποχρέωση της επιχείρησης όπως αλλού το κράτος το κράτος απευθείας παρέσχε σε όλες τις επιχειρήσεις σε όλες τις γυναίκες αυτή την, ε, την ευκολία για τη φύλαξη των παιδιών ε, απλώς είναι τα πράγματα περίπλοκα Κάναμε μια μελέτη για, για τους το πυρητικό προσωπικό μας στο σπίτι και τελικά περισσότερες συνομιλίες στην Ισπανία. Έχουν εισαγάγει η Ισπανία εκατομμύρια μεταναστών για να βοηθούν να καθαρίσουν το σπίτι και μετά... Αυτά για τις οικιακές βοηθούς. I have a disadvantage because probably something, uh, something I miss. Uh. Α, υπάρχει κάτι ίσως που δεν ε, κατάλαβα, δεν πέρασα από τη μετάφραση, δεν ξέρω. The outcome of the translation was that uh, uh in... Αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι στην Ισπανία η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας επιδεινώνεται. Δεν ξέρω, αυτό, αυτό, ήταν, αυτό, αυτό ρωτήσατε. Would θα θέλατε, λέει πρόεδρος, να μας το εξηγήσετε. Δημοσιογράφος. Είπαμε ότι έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στην υγεία, την παιδεία, για παράδειγμα τώρα έχει γίνει μεγάλη περικοπή στους, στους, για τους δάσκαλους και καθηγητές. Και αυτό οδήγησε στο πολλές γυναίκες οι οποίες εργαζόντουσαν σε κάποια ας πούμε επιχείρηση, σε κάποια εταιρεία ξαφνικά χτυπήθηκαν από την κρίση. Και τώρα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό που δεν κάνουν οι, οι άντρε. Δηλαδή τη δουλειά στην οικογένεια, το σπίτι κλπ. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Yes, of course. Uh, uh, what we are... Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Λέμε το τι θα κάνουμε όσον αφορά το, το, το, το, θέμα που συζητάμε σήμερα στο μέλλον, ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Κάθε, κάθε κρίση έχει την αρχή και το τέλος της. Είναι αδύνατον. Κανείς να όλα, τα καλύψει όλα, όλα, όλα τα, τα κακά που φέρνει η κρίση ούτε καν μπορώ να καλύψω το ερώτημά σας 100% γιατί τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεσμενή για τις γυναίκες. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι το δεύτερο κύμα των μέτρων λιτότητας είχε ακόμα τις επιπτώσεις για τις γυναίκες παρά για τους άντρες. Στο πρώτο κύμα μέτρων επλήγει η βιομηχανία, ο οικονομικός τομέας, οπότε όντως τότε είχαμε δυσμενή αποτέλεσματα για τους άντρες. Όμως τώρα τα σχετικά μέτρα επέδρασαν πολύ χειρότερα για τις γυναίκες. Το θέμα όμω σηκώνει συζήτηση. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα πρέπει κάπως να ολοκληρώσουμε. Ε, ήρθε τώρα ο πρόεδρο μας, ο όμως, για να δούμε. Έχουμε ένα ερώτημα και κατόπιν ε, οι υπόλοιποι τρει του πάνελ να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εστονικά, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία. Μπάρμπαλ λέγεται η εφημερίδα μου και θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα προς την κυρία Χόκκιν. Δύο μάλλον. Πρώτον, τι θα μπορούσατε να μας συστήσετε ως μέτρο ε, για, στην Εστονία. Έχουμε μία μισθολογική διαφορά 30%. Λέτε ότι δεν βοηθάει η εκπαίδευση. Μας λέτε ότι τα νέα νομοσχέδια σίγουρα δεν θα φέρουν την αλλαγή. Ωραία, τι προτείνετε λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα τόσο πολύ καιρό που θα εκτιμούσα αν μου λέγατε τι πιστεύετε για τις ποσοστώσεις ε, στις διευθυντικές θέσεις των επιχειρήσεων. Θέλετε όλοι να πείτε κάτι. Ωραία. Η μία μετά την άλλη και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τους διάφορους παράγοντες ε, και, αυτού και κυρίως να ασχοληθούμε με αυτούς που μπορούμε να ρυθμίσουμε ο πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα που εξαρτάται από τα κράτη, είναι εθνική αρμοδιότητας θέματος όπως τα ωράρια ε, στα σχολικά, στη Γερμανία ας πούμε πολλές φορές εξαρτάται και από το κρατήδιο. Το θέμα είναι βέβαια να δούμε εδώ γιατί θέσεις απασχόλησης υποβάλλουν υποψηφιότητες οι άντρες και οι γυναίκες. Και αν η αντιμετώπιση, οι συνθήκες και ο μισθός βεβαίω και οι αποδοχές είναι αντίστοιχες και ίσες. Και το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτές τις ε, θέσεις για να συγκρίνει και τις αποδοχές, γιατί μπορούμε να το πάμε και πιο πέρα αυτό το σημείο σύγκρισης και να αναρωτηθούμε αν μια δασκάλα δημοτικού έχει λιγότερο επίπονη εργασία από κάποιον που ε, είναι βαθμό στέλεχο μιας επιχείρησης με αποδοχές που δεν συγκρίνονται. Στην ε, Γερμανία βλέπουμε λοιπόν ακόμα και μεταξύ των κρατηδίων να υπάρχουν διαφορές. Σε εμά, όπως ξέρετε, υπάρχει το ομοσπονδιακό κράτος και υπάρχει και το επίπεδο του κρατηδίου. Και τα θέματα αυτά ρυθμίζονται σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά επαναλαμβάνω και εγώ ότι πέραν του εθνικού επίπεδου υπάρχει ίσως και το ευρωπαϊκό που μπορεί να δώσει κάποια κίνητρα, κάποια όθηση και μετά βεβαίως είναι το μεγάλο θέμα της εφαρμογής, της υλοποίησης. Πώς δηλαδή όλα αυτά τα νομοθετικά κείμενα θα γίνουν πραγματικότητα. Πώς θα υλοποιηθούν τι δυνατότητες υπάρχουν προσφυγής, τι δυνατότητες ενημέρωσης για να ξέρουν οι γυναίκες στα διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουν αυτές τις δυνατότητες. Και βεβαίως θα πρέπει το κοινοτικό δίκαιο να μεταφερθεί κατόπιν να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και να γίνει πραγματικότητα για τους πολίτες της Ευρώπης. Ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι γυναίκες αυτά τα επαγγέλματα και όχι τα άλλα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υπεύθυνε μόνο οι γυναίκες. Και αυτό ξεκινάει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήδη στα σχολεία υπάρχουν οι μέρες όπου τα αγόρια και κατόπιν τα κορίτσια σε διαφορετικές μέρες γνωρίζουν τα διάφορα επαγγέλματα με σκοπό να διαλέξουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η ανατροφή των παιδιών το πώς τους κατευθύνουμε. Τι είναι σημαντικό για μας. Η ανατροφή των παιδιών μας με αξιοπρέπεια. Και βεβαίως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση μια γυναίκα να επιλέξει ένα επάγγελμα όπως παραδείγματο χάρη μηχανικός επειδή είναι ένα καλοπληρωμένο επάγγελμα να εγκαταλείψει κάτι που της αρέσει το οποίο όμως είναι χαμηλό στο επάγγελμα ε, ακριβώς αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ναι, εγώ είμαι υπέρ των ποσοστώσεων, να απαντήσω και σε αυτό. Σε εμά είχε αποτέλεσμα. Και βεβαίως είμαστε υπέρ των ποσοστώσεων. Το αποτέλεσμα βεβαίως δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών μας. Το ερώτημα για τις ποσοστώσεις και εγώ μπορώ να απαντήσω. Είμαστε υπέρ, είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα για να μην υπάρχουν οπισθοχωρήσεις. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που μου φαίνεται πολύ σημαντικό και θα τελειώσω με την δική μου παρουσίαση. Όλα όσα ζούμε αυτές τις ημέρες, πολιτική λιτότητας, πακέτα για την Ελλάδα, μέτρα για την Ισπανία ή αλλού, Όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραγωγικά και να οδηγήσουν σε οπισθοχώρηση για όλους αυτούς τους τομείς που συζητούμε σήμερα. Θέλουμε να μειωθούν οι κίνδυνοι να πέσουν οι γυναίκες στη φτώχεια, να βρίσκονται διαρκώς στις πιο χαμηλόμιστες κατηγορίες. Θέλουμε να μειωθεί το χάσμα των μισθών και των αποδοχών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Και θέλουμε να μπορούν οι γυναίκες να έχουν δυνατότητες και υπηρεσίες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, παραδείγματος χάρη. Να φύγουμε από τα παλιά κλισέ του καταμερισμού των ρόλων και των επαγγελμάτων και αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα, μείωση του χάσματος μισθών που υπάρχει μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Η κυρία Χάκεμ, σύντομα σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε. Δεν είμαι υπέρ των ποσοστώσεων. Απλώς θεωρώ ότι ε, ορισμένες φορές οι αλλαγές γίνονται πιο αργά από ό,τι περιμένουμε και γίνεται, γίνονται οι αλλαγές ε, παρότι δεν είναι τόσο ραγδαίες όσο θα επιθυμούσαμε. Νομίζω ότι θα υπόλοιπα αν υιοθετήσουμε τις ποσοστώσεις ε, ε, και σας παραπέμπω στην έκθεσή μου. Σχετικά με το 30% την μισθολογική διαφορά στην Εστονία. Ε, μου κάνατε μία ερώτηση. Θα ήθελα εγώ να ξέρω πώ αιτιολογείται αυτό, διότι όπω ε, είδα στη μελέτη μου σε σχέση με του ε, φαρμακοποιού, δεν τίθεται ζήτημα διακριτική μεταχείρισης ή ίση αμοιβή. Σχετίζεται, όπω σα έλεγα, με τι επιλογέ που κάνουν οι γυναίκε αν σε εθελοντική βάση επιλέγουν κάποιε συγκεκριμένε δουλειέ ή πιο περιορισμένο ωράριο απασχόληση Είναι δική του επιλογή και α αρχίσουμε να προσποιούμαστε ε, επιτέλους ε, ότι υποφέρουμε ε, προβάλλοντας τους λανθασμένους λόγους. Ξέρετε υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, έχουν, που εργάζονται πάρα πολλές ώρες, πρέπει να πηγαίνουν επιχειρηματικά ταξίδια, αυτό δεν το θέλουν οι περισσότερες γυναίκες, έχουν περισσότερο άγχος κτλ. κτλ. Ξέρετε υπάρχουν λόγοι για τους οποίους επιλέγουν τις δουλειές που επιλέγουν έχουν γυναίκες. Ε, είναι προβλέψιμο το άθος εργασίας, ε, ε, φυσιολογικά ωράρια, αποδίνει μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε θα πρέπει να δούμε το συνολικό πακέτο, δηλαδή πώς αμείβεται η δουλειά, αλλά όχι μόνο τι, προ... τι απαιτεί μία δουλειά. Ε, και ξέρετε υπάρχουν και άλλες θέσεις εργασίας με χαμηλή αμοιβή αλλά που είναι, ε, παρουσιάζουν άλλα θέλγητρα όπως σας έλεγα προβλεπόμενα ωράρια, ε, καλή όρια απασχόλησης, καλός εργοδότης κτλ. Δηλαδή θα πρέπει να δείτε πώς εξηγείται αυτό το 30% και ενδέχεται να μην συνιστά πρόβλημα αυτό που νομίζετε ότι ευθύνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χακίν, λέει η κυρία Κόχ Κυρία Τόμσεν, θέλετε να κάνετε και μια τελευταία παρατήρηση και θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρό μα. Ε, ευχαριστώ. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω ε, ταξίδια. Πήγα στη Βραζιλία τι προάλλε. Ε, μ' αρέσει να πετάω στην πρώτη θέση. Πολλά μου αρέσουν. Και οι φίλε μου μου λένε ότι και εκείνες θα ήθελαν αλλά δεν είχαν τις ευκαιρίες να το πετύχουν όπως το είχαν σχεδιάσει, διότι ε, στην Ευρώπη υπάρχει μία ε, οροφή που δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να υπερβούμε. Δεν έχουν όλες τις ίδιες ευκαιρίες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν και οι δυνατότητες εκλογής που έχουν οι άντρες επιλογής και πολλές φορές Μπορεί κάποιος να πει ότι μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα νηπιαγωγείο όλη την ημέρα παίζει. Τι δουλειά είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις συνεισφορές σας, ε, για τις ιδέες σας. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος μας είναι άντρας. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το Ευρωμαρόμετρο. So, we, we arrive at the end of our... Φτάνουμε σίγουρα στο τέλος του προγράμματός μας. Όπως είπε η κυρία Κό. Προεδρεύει τώρα ένας άντρας. Για πρώτη φορά σήμερα. He is the, the, the chair of the είστε πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών. Θα παρουσιάσετε το Ευρωβαρόμετρο που θα δημοσιευθεί σήμερα. Η γάμα θέλετε επικοινωνία, ε, ζήτησε το Ευρωβαρόμετρο και θέλετε κι εσείς να πείτε κάποια λόγια, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Γκούσταψον για να μας παρουσιάσει τη μελέτη, θα ήθελα να διευκρινίσω δύο-τρία τεχνικά ζητήματα. Αυτό το ευρωβαρόμετρο διεξήχθη από την Tennis Opinion στον Ιανουάριο του 2011 καλύπτει τα 27 κράτη, ε, περίπου 27.000 Ευρωπαίοι πάνω από 15 χρονών ρωτήθηκαν τηλεφωνικά με στόχο να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την ε, έλλειψη ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Επίσης, ο στόχος ήταν να ασχοληθούμε όλος ιδιαίτερος με τις μισθολογικές διαφορές. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Αν δεν ομιλείτε τη Σουηδική, βάλτε τα ακουστικά σας. Ja, Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχω την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω αυτή τη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου ε, σχεδόν 27.000 Ευρωπαίοι εξέφρασαν την άποψή τους ε, και θα ήθελα να αρχίσω κάνοντας μια γενική παρουσίαση σχετικά με τις ε, ανισότητες. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην πρώτη σελίδα που περιγράφει την κατάσταση, όπως βλέπετε στον πίνακα σχετικά με τις απόψεις αυτών των ανθρώπων που μας δείχνουν ότι ε, κατά πόσο μάλλον είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα. 50% πιστεύουν ότι είναι σημαντικά τα ζητήματα ανισότητας των δύο ε, ε ένα στου δύο δηλαδή πιστεύει ότι είναι σημαντικό το ζήτημα. Εγώ ήλπιζα ω πρόεδρο τη Επιτροπή Γυναικών θα ήταν κάπω υψηλότερο το ποσοστό, διότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι γυναικείο ζήτημα το ζήτημα τη ισότητα των δύο φύλων. Είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε θα έπρεπε να είναι υψηλότερο το ποσοστό, όχι μόνο εμεί σίγουρα πιστεύουν ότι είναι σημαντικό. Τέλο πάντων, ε, ίσω είναι και καλό. Αυτό θα δούμε. Επόμενη σελίδα. Ε, κατανομή, βλέπετε τι στις διάφορες χώρες, την κατανομή αναχώρα και υπάρχουν μεγάλες διαφορές όπως παρατηρείτε σχετικά με τις απαντήσεις. Η Ισπανία, η Γαλλία και η Ρουμανία είναι στην κορυφή του καταλόγου και κάτω-κάτω είναι η Βουλγαρία, η Φινλανδία και η Εστονία. Παρακαλώ επόμενη διαφάνεια. Σε αυτή τη σελίδα τίθεται το ερώτημα ε, τι έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Ε, οι πώς οι ερωτηθέντες ε, αντιλαμβάνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το τομέα. 60% λοιπόν των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Πολύ καλό αυτό βεβαίως. Ε. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί από πού ξεκινήσαμε σε κάθε χώρα. Όντως υπήρξε βελτίωση, αλλά από πού ξεκινήσαμε. Στη συνέχεια, αρχίζουμε με την κατανομή, βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, όλοι οι ερωτηθέντες από όλα τα κράτη-μέλη, ε, θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό είναι θετικό. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε ένα πίνακα που πρέπει να δούμε προσεκτικά. Ε, μας δίνει πολλές πληροφορίες, εγώ θα ασχοληθώ μόνο με δύο πτυχές. Πρώτον, με σαφήνεια, αν εξετάσουμε πώς απαντούν οι άντρες και οι γυναίκες σχετικά με το αν είναι σημαντικό το θέμα της ισότητας ή όχι, βλέπουμε ότι έχουμε με ισοψηφία 50-50 σχεδόν, λίγο λιγότεροι οι άντρες, ε, ε, εντάξει, δεν σας ξαφνιάζει αυτό, φαντάζομαι. Άλλοι πάλι ε, μας είπαν ότι όσο νεότερος είναι κάποιος, τόσο ε, λιγότερο σημαντικό θεωρεί ότι είναι το ζήτημα της ισότητας ε, ε, των δύο φύλων. Δηλαδή, όταν, όσο ζει κανείς και μεγαλώνει, αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια και συνειδητοποιεί ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, όντως δεν έχουν ίση αμοιβή οι γυναίκες, είναι εκτεθειμένες στη βία, έχουν χειρότερους όρους εργασίας, ε, είναι λογικό σε πιο προχωρημένη ηλικία να συνειδητοποιεί κανεί τα προβλήματα. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα και βλέπουμε ε, την επόμενη ερώτηση. Κατά την άποψή σας, ε, λέει η ερώτηση, από στον τομέα της ισότητας ποια είναι τα τρία πλέον σημαντικά θέματα. Με σαφήνεια φαίνεται από τις απαντήσεις ότι το βασικότερο ζήτημα είναι η βία των ανδρών κατά των γυναικών. Ε, στη συνέχεια μισθολογικό χάσμα και στην τρίτη θέση ε, η πορνεία και η εμπορία ανθρώπων. Στη συνέχεια βλέπουμε την επόμενη ερώτηση ποιο είναι το σημαντικότερο ε, θέμα. Και βλέπετε ε, ότι έχετε ε, τις δύο τις δύο, τα δύο χρώματα, το μπλε και το κίτρινο και βλέπετε ότι οι τάσεις είναι παρόμοιες. Συνδυάζονται δηλαδή αυτά τα δύο ερωτήματα, γενική επισκόπηση ε, και η πιο συγκεκριμένη σχετικά με την ανισότητα των δύο φίλων. Να δούμε τώρα το θέμα της εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων κατά τη διαστολή με την εκπροσώπηση στον πολιτικό βίο. Ξαφνιάστηκαν με τα αποτελέσματα ε, γιατί είναι υψηλότερα τα ποσοστά τις επιχειρήσεις από ότι ε, σε πολιτικά, θεσμικά όργανα, πολιτικό, πολιτικού χαρακτήρα. Κανονικά τα όργανα της δημοκρατίας πρέπει να εκπροσωπούν ορθότερα το λαό και άρα θα έπρεπε να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την εκπροσώπηση των γυναικών. Όταν μιλάμε δηλαδή για κοινοβούλια που εκπροσωπούν κατεξοχήν ε, τους πολίτες, βλέπουμε ότι εκεί είναι υψηλότερα τα ποσοστά σε σχέση με τις επιχειρήσεις και μπορούμε έτσι να περάσουμε στην επόμενη σελίδα. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με το ποιο είναι το σημαντικότερο ζήτημα. 12% ε, θεωρούν ότι το σημαντικότερο είναι η βία. Παρακαλώ, δείξτε μου και την επόμενη διαφάνεια. Στη συνέχεια σας είπα, δεύτερη θέση είναι, ε, στη δεύτερη θέση είναι η μισθολογική διαφορά Υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, ανάμεσα στην αντίληψη αναχώρα σχετικά με το ποιο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στον τομέα της ε, καταπολέμησης των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ε, μεγάλο πρόβλημα η μισθολογική διαφορά, ναι ή όχι. Εδώ βλέπουμε σχεδόν 7 από τους 10 θεωρούν ότι όντως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και είναι ενδιαφέρον γιατί μόνο 50% ισχυρίζονται ότι είναι σημαντικό το ζήτημα της ισότητας αλλά όταν περνάμε στη μισθολογική διαφορά ανεβαίνει το ποσοστό στα 70%. Είναι συναρπαστικά τα αποτελέσματα αυτού του ευρωβαρόμετρου. Επίσης, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία είναι υψηλά τα ποσοστά, θεωρούν ότι είναι σημαντικό το ζήτημα της ε, μισθολογικής ε, διαφοράς. Μάλτα, Λιθουανία, Λετωνία είναι αυτοί που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά, αν βλέπω καλά. Επόμενη σελίδα. Please go back. Sorry. Ε, συγγνώμη την προηγούμενη θέλω, όχι την επόμενη, ζητώ συγγνώμη. Είμαι γρήγορος, δεν λέω, αλλά τόσο γρήγορος δεν είμαι. Ωραία. Για να δούμε, σε αυτή τη διαφάνεια, ε, ποια είναι η ερώτηση. Πάλι έχουμε το θέμα της μισθολογικής διαφοράς, πόσοι πιστεύουν ότι είναι το πιο σημαντικό και βλέπουμε τις απαντήσεις αναφύλλω. για αυτό το ζήτημα. Με σαφήνεια προκύπτει από τους ε, ε, ερωτηθέντες ε, ότι ακόμη και οι άντρες σε ποσοστό 62% θεωρούν ότι είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που θεωρούν ότι είναι σημαντικό λοιπόν ε, το ζήτημα της μισθολογικής ε, διαφοράς. Ε, στη συνέχεια βλέπετε το θέμα της ηλικίας που σχολίαζα νωρίτερα, δηλαδή όσο νεότερος είναι κάποιος τόσο λιγότερο θεωρεί ότι είναι σημαντικό το θέμα της διαφοράς ανάμεσα στα δύο φύλλα. Συνεχίζουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εντοπίζονται. πώς έχει ερώτηση τώρα. Αν ξέρουμε ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά στη τάξη του 17,5%, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το καταπολεμήσουμε, Πώς ρωτήθηκαν όλοι πρέπει να ρυθμιστεί το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο. Οι περισσότεροι είπαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 38% σε εθνικό επίπεδο και το τοπικό επίπεδο ήταν στα 11%. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρέπει να επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση του ζητήματος. Κάτω περνούμε στο επόμενο ερώτημα. Με πώς, με νομοθετικά μέτρα, με συστάσεις, με αποφάσεις, ε, με ποιο τρόπο. Ε, βλέπουμε στη συνέχεια την κατανομή αναχώρα και αυτούς, αυτές οι χώρες που είναι στα αριστερά θεωρούν ότι το σημαντικότερο επίπεδο που μπορούμε κάτι να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση είναι το ευρωπαϊκό. Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο είναι πάνω-πάνω και στη συνέχεια έχουμε από την αντίθετη πλευρά Τσεχία, Εστονία, Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά. På ε, στην επόμενη σελίδα βλέπουμε ότι ερωτήθηκαν οι πολίτες σε ποια μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλλουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να μειωθεί η μισθολογική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Ε, εδώ δεν υπάρχει σαφής ε, διαχωρισμός απόψεων. 27% μόνο θεωρούν ότι ε, πρέπει ε, να εγκρίνουμε αυτά τα μέτρα για διευκόλυνση τη πρόσβαση στην αγορά εργασία. 26% ε, θεωρούν ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσει. άλλοι ένα άλλο, εγώ πιστεύω ότι το 26% θα ήταν υπέρ των ήπιων μέτρων, δηλαδή να ενθαρρύνουμε, να τονώσουμε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην αγορά και όχι να τιμωρήσουμε στη συνέχεια. Όταν διαβάζω εγώ αυτά τα αποτελέσματα, συνειδητοποιώ ότι μπορούν να κρύβονται πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτά τα στοιχεία, ε, διότι ε, όταν γίνεται μια δημοσκόπηση, δεν καταλαβαίνω ερωτηθέντες ακριβώς όλες τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν. Ε. Ε, αναφέρομαι στους υπόλοιπους παράγοντες που διαμορφώνουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας και που μπορούν να επηρεάσουν τις διαφορές. Όπως έλεγε η κυρία Μπάουερ, παραδείγματος χάρη θέματα πατρικής ε, άδειας, ε, ε, γονικής άδειας, ποιο ποσοστό από τον μισθό χρησιμοποιείται για το σπίτι, πώς πώς επηρεάζεται η επιλογή των γυναικών αν θα κάτσουν στο σπίτι, δηλαδή για να φροντίζουν τα παιδιά τους ή όχι, ανάλογα με το πόσα χρήματα βγάζουν, αν είναι υψηλότερος ο μισθός τους, χαμηλότερος σε σχέση με το άντρα τους κτλ. Στη συνέχεια, βλέπουμε και πάλι ε, τα ίδια ποσοστά μπορούμε να περάσουμε αυτή τη διαφάνεια ακόμη και την επόμενη και φτάνουμε στην τελευταία εικόνα με, με ηλικιώδη ταχύτητα φτάσαμε στο τέλος. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο σημαντικό να προσθέσω. Δεν θέλω να δαπανίσω άλλο το χρόνο σας, οπότε Υπάρχουν ερωτήσεις? Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για λίγες ερωτήσεις. Ε, παρά το ότι έχουμε βγει λίγο από το χρόνο μας. Διακρίνω. Κάποιον από το προηγούμενο πάνελ να θέλει κάτι να ερωτήσει. Παρακαλώ. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω το ότι αυτό το οποίο ρωτήσατε, το, είχε και το Σλατή, 17,5% είναι η διαφορά στο μισθολογικό χάσμα. Αυτή, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, λέει ο μιλητή. Δεν έλεγαν αυτό όμω τα στατιστικά. Είπαμε ότι για όλα τα επαγγέλματα ο μέσος μισθός του ενός και του άλλου. Άρα δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω εδώ, απλώ παρουσιάζω τα αποτελέσματα. Δεν φταίω εγώ. Ίσως ε, μπορεί να σας διευκρινίσει ο συνάδελφο. Έτσι όπως ε, τίθεται το ερώτημα δεν είναι ειλικρινέ, γιατί αυτό που σας λέω είναι το, το, το στοιχείο, το πραγματικό περιστατικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτά ερωτήσεις μέσω του Ευρωβαρόμετρου που είναι παραπλανητικές, ανηλικρινεί, αυτό είναι τρομερό. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο ως κοινωνιολόγος, επιστήμονα, πρόεδρος. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται. Δεν κατάλαβα γιατί είναι λάθος. Δεν είναι αυτό. Το μισθολογικό χάσμα στις στατιστικές αφορά όλο το εργατικό δυναμικό και όχι επί τη βάση της δουλειάς ε, ίσης αξίας Α, αυτό είναι τελείο πρόεδρος, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, πρόκειται για μέσο όρο. Αυτό συγκρίνουμε. Δεν είναι. Δεν είναι η αξία. Είναι απλώς ένα πραγματικό περιστατικό. Αυτό εννοείται. Η ερωτώσα. Η ερώτηση είναι ανηλικρινής 100%. Πρόεδρος. Η ερώτηση ήταν ποιες ανισότητες μεταξύ των φύλων θεωρείται ότι είναι οι πιο μεγάλες. Ο κύριος το Κοιτάξτε, μας αυτά τα στοιχεία μας έδωσαν κυρία μου όταν ε, συντάξαμε το ερωτηματολόγιο το 17,5%. Ε, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σε συνεργασία με την ε, γραμματεία της Επιτροπής Γυναικών. Οπότε μας έδωσαν αυτό το στοιχείο όπως ε, πρόκειται για την ε, ε, μισθολογική διαφορά γυναικών ανδρών. Αυτά μας έδωσαν. Μα, απάντηση. Ισχύει αυτό το αριθμητικό στοιχείο, αλλά είναι για όλη την αγορά εργασίας, όχι για αμοιβή, για την ίδια δουλειά. Ε, όταν δεν υπάρχει ίδια αμοιβή για ακριβώς την ίδια δουλειά, εκεί σε αυτό έγκυται η διακριτική μεταχείριση, ενώ εσείς χρησιμοποιείτε ένα ποσοστό που ισχύει σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Ανεξαρτήτως ε, παροχής υπηρεσιών, ε, απάντηση, νομίζω ότι πρόκειται για πρόβλημα μεθοδολογίας. Yeah. Uh, I, I take that in Swedish, it's θα μιλήσω σου ειδικά, γιατί είναι ευκολότερο για μένα. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά δεν είναι ότι κάποιος προσπάθησε να εξαπατήσει τους άλλους και εμένα προς Θεού. Εννοείται ότι το 17,5% είναι ε, ε, ευσταθή, αυτό καθε αυτό, αλλά είναι το, ε, σχετίζεται με το σύνολο του μισθού ε, και όχι για την ίδια δουλειά, ίδια αμοιβή, αυτή την αρχή που σχολιάσαμε. Κοιτάξτε, να, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εντελώς παραπλανητικών στοιχείων που προκύπτουν από μελέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι, λυπάμαι. Mm, I Δεν ξέρω. Προεδρεύουσα, δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο, κάποιος άλλος θα κάτι να ρωτήσει, δεν ξέρω. Όχι, Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο πριν τελειώσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ε, μια αξιολόγηση έξωθεν αν ευσταθούν δεν ευσταθούν τα στοιχεία. Δεν μπορείτε ε, ίσως να δυσφημείται όλα τα αποτελέσματα της έκθεσης. Μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό το ερώτημα, αλλά ξέρετε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βλέπει κανείς τα ζητήματα ε, ανισότητας. Ε, εάν θεωρείτε ότι δεν ισχύει αυτό το ερώτημα να το αφαιρέσουμε, αλλά όχι να απαξιώσετε ολόκληρο το ευρωβαρόμετρο θα πρέπει ε, ε, βεβαίω να ενημερωθώ πρωτού αποφασίσουμε τίποτα, ε, γιατί δεν γίνεται αλλιώ να πάρουμε αποφάσει. Κοιτάξτε, το, ο στόχο του Ευρωβαρόμετρου ο ίδιο είναι να παραπλανηθούν οι ερωτηθέντε. Δηλαδή, του λέτε ότι είναι πρόβλημα η μισθολογική διαφορά. Ναι, αλλά μιλάμε για μισθολογική διαφορά για την ίδια δουλειά, όχι γενικά. Λοιπόν, οι ερωτήσει, οι απαντήσει εδόθησαν διότι θέσατε το ερώτημα με παραπλανητικό τρόπο πω Πώς έγινε, ποιος το έκανε, δεν ξέρω, πάντως έγινε και απαξιώνεται από μόνο του το ευρωβαρόμετρο ε, και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που νομίζετε ούτε όπως μας τα παρουσιάσατε. Δεν ισχύει αυτό, ε, το αποτέλεσμα όπως μας το παρουσιάσατε. Ε, δεν μπορείτε επίσης να τα ρίχνετε όλα κατά το χαλί, να λέτε ότι είναι μεθοδολογικό ζήτημα. Πολιτικό είναι πώς παρουσιάζεται το ευρωβαρόμετρο, πώς θα αντιμετωπίσουμε πώς το παρουσιάζουμε. Είναι αν και παραπλανητικές οι ερωτήσεις και δείχνουν ότι η μισθολογική διαφορά είναι πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει. Εάν όμως μιλούσαμε για ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά, θα είχαμε διαφορετικέ απαντήσει. Μιλάτε γενικά εδώ για την μισθολογική διαφορά που δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτό που μα ενδιαφέρει να μελετήσουμε, δεν έχει γίνει προσαρμογή. Γι' αυτό απαξιώνεται ολόκληρη, ολόκληρη μελέτη. Συγγνώμη, θα ακούσουμε τον πρόεδρο. Ξέρετε, θα δημιουργηθούν εξίσου πολλά προβλήματα με αυτό που κάνετε τώρα. Το ίδιο κάνετε κι εσείς λοιπόν. Ε, Απαξιώνει το ολόκληρο το ευρωβαρόμετρο. Είπαμε, υπάρχει ένα πρόβλημα, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε ολόκληρη την έκθεση. Πρέπει να συνυπολογίσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία και όχι να απαξιώσουμε ε, το, ολόκληρη τη μελέτη επειδή υπάρχει ένα μόνο ε, πρόβλημα. Δεν γίνεται ούτε από επιστημονικής πλευράς. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα ατυχές, θα το πω έτσι, ερώτημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, είναι παράλογα όλα τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ παράξενο που ε, τηρείται αυτή τη στάση και αυτή είναι πολιτική στάση που τηρείται. Νομίζω με παρανοήσατε. Εάν ρωτήσετε κάποιο, είναι κακό πράγμα ο φόνο, όλοι θα πούνε ναι, ναι, κακό είναι. Αν στη συνέχεια κάνετε άλλε ερωτήσει, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα με τι πολιτικέ ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο και ούτω καθεξή θα πάρετε τις απαντήσεις. Αλλά απλώ λέω ότι αν το εφαλτήριο είναι λανθασμένο, δηλαδή αρχίσετε με το φόνο, ε, λοιπόν, όλη η μελέτη θα βασιστεί σε αυτό. Δεν είναι μία ερώτηση, είναι η ερώτηση που καθορίζει όλο το, όλη την υπόλοιπη μελέτη. Είναι, είναι πλημελής η πληροφορία, είναι παραπλανητική, καταλαβαίνετε, και να λέμε μετά... Ε, ζητώ συγγνώμη σα διακόπτω, διότι δεν ήταν η μελέτη όλη για την μισθολογική διαφορά, ήταν για τις ανισότητες και τα ερωτήματα που ε, ετέθησαν σχετίζονταν με τη μισθολογική διαφορά. Ε, πώς ήταν η ερώτηση, εσείς ε, πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι η μισθολογική διαφορά. Αυτή ήταν η ερώτηση και ήταν ελεύθεροι οι πολίτες να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη, δηλαδή κατά τη δική τους άποψη ποια είναι η βασικότερη ανησυχία, το βασικό το πρόβλημα για τις γυναίκες. Κάποιοι είπαν ότι είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα γενικότερα, κάποιοι αναφέρθηκαν στη μισθολογική διαφορά, ζητώ Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα αυτή την άγουσα. Και, ε, είναι μεθοδολογικό το πρόβλημα. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, άλλες ερωτήσεις. Νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε εδώ. Άντε, άλλη μία τελευταία. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι αυτό για την βία των ανδρών κατά των γυναικών. Υπάρχει κάποια χώρα που θεωρεί ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα ανισότητας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη βία των γυναικών σε αυτή τη χώρα ή σημαίνει ότι σε εκείνη τη χώρα οι, οι, πολίτες ε, έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του προβλήματος από αλλού ή και τα δύο. Πρόεδρος. έχετε. Δεν μπορούμε ε, να που ισχυριστούμε ότι επειδή είναι υψηλό ποσοστό σε μια χώρα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην άλλη. Ξέρετε, το υψηλό ποσοστό μπορεί να σημαίνει αυξημένη συνειδητοποίηση του προβλήματο. Άρα φαίνεται περισσότερο για άποψη αυτή τη χώρα. Υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να δούμε προσεκτικά αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο. Υπάρχουν διάφορε συνιστώσει που εξηγούν το ποσοστό των απαντήσεων και τι ίδιε απαντήσει. εκτός μικροφώνου. Φτάνουμε στο τέλος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχετε το ευρωβαρόμετρο και σε χαρτί και διαδικτυακά ε, έχετε το αρχείο. Θα σας στείλουμε το αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα έχετε άπλετο χρόνο να μελετήσετε τα ζητήματα. Αν έχετε ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία μπορείτε να τα διαβάσετε στη γραμματεία και θα σας απαντήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πρόεδρε, ε, για την συμμετοχή σας, για την παρουσίαση του Ευρωβαρόμετρου. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Ε, όπως ε, κάποιες πρακτικές ε, πληροφορίες, όπως σας είπα, μπορεί είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε στη συνεδρίαση των Εθνικών Κοινοβουλίων που διοργανώνει η Επιτροπή των Γυναικών αύριο. Εκεί θα συζητήσουμε το ίδιο θέμα με βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και με εμπειρογνώμενες. Στις 7 σήμερα το βράδυ έχουμε την Begenham, μια ταινία που προβάλλει η Επιτροπή των Γυναικών, μια μέρα στον Τάγκενχαμ ε, και δεν ξέρω αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, πάντως είστε καλεσμένοι. Επίσης, ε, αυτή τη στιγμή στο δεύτερο όροφο, όχι εδώ, θα ανέβετε έναν όροφο, ε, υπάρχει μια δεξίωση και έκθεση στον ίδιο όροφο και εκεί είστε καλεσμένοι. Θα στείλουμε τις εκθέσεις και θα γίνει το follow-up, όπως είπαμε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η τόσο εντατική ημέρα ε, και περιμένουμε παρατηρήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς, ε, γιατί εργάστηκαν σκληρά. Καλό βράδυ.